Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ξεκινάμε συνάδελφοι. Je remercie le Lewandowski. Ευχαριστώ τον κύριο Λεβαντόσκι, τον χαιρετώ, αυτόν και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με ό,τι συνήθως κάνουμε, ο Επίτροπος έρχεται να μας παρουσιάσει πριν από οπουδήποτε αλλού στην Επιτροπή μας το προσχέδιο για το 2014 το οποίο σήμερα το πρωί υιοθέτησε το σύνολο των επιτρόπων. Πρόκειται για μια έκτακτη συνεδρίαση αυτή που έχουμε εδώ σήμερα. Σας υπενθυμίζω ότι θα έχουμε την τακτική μας προγραμματισμένη συνεδρίαση αύριο το πρωί στις 9. Και σας ενημερώνω επίσης ότι ζήτησα ήδη από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να οργανώσει μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας την επόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο στις 6.30. Αυτό το είχαμε ζητήσει χρονικά θα έλεγα για τους συντονιστές τη στιγμή αυτή τη χρονική αλλά θα είναι μια δημόσια και ελπίζω μια ολομέλεια της Επιτροπής μας για να δούμε ακριβώς που βρισκόμαστε σε σχέση με το πολιετές πλαίσιο που δεν θα συζητήσουμε σήμερα, το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει και κλεισμένο των θυρών τη Δευτέρα και στο οποίο θα πρέπει να επανέλθουμε πριν από την ψηφοφορία η οποία πιθανώς να ε, ε, γίνει, να ζητηθεί να γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλειά μας. Είδατε λοιπόν την ημερήσια διάταξη, δεν έχουμε κάτι άλλο στην ημερήσια διάταξη εκτός από την παρουσίαση. Η παρουσίαση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω τον ε, λόγο αμέσως στον Επίτροπο Λεβαντόσκι. Thank you. Good morning. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο στάδιο του πρώτου προϋπολογισμού μέσα στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και είναι ένας προϋπολογισμός για 28 χώρες, όχι 27, αλλά 28. Τα καλά νέα είναι ότι σήμερα το πρωί η Κόρεπελ συμφώνησε για την Κροατία. Αυτό είναι ουσιαστικό. Μπορούμε να καλωσορίσουμε ένα ακόμα μέλος μιας οικογένειας 28 μελών πια. Όπως φαίνεται λοιπόν στην πρώτη διαφάνεια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ξεκινούμε χωρίς ένα συμπεφωνημένο πλαίσιο δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά σεβόμαστε όλους τους κανόνες ότι δηλαδή μετά την επίσημη έγκριση του προϋπολογισμού θα παρουσιάσουμε ε, θα, ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε τον προϋπολογισμό εγκαίρως ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει του άρθρου 314 είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε προβλέψεις σε όλες τις γλώσσες πριν από την 1η Ιουλίου και το σχέδιο προϋπολογισμού, το προσχέδιο μέχρι την 1η Ιουλίου και το σχέδιο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Σε φυσιολογικές συνθήκες ακολουθούμε μία πραγματιστική προσέγγιση. Ήδη παρουσιάζουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού στο τέλος Απριλίου και αυτό δίνει περισσότερο χρόνο και για το, και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο για, για τις αναγνώσεις, τη διαδικασία των αναγνώσεων του προϋπολογισμού. Μπορούμε όμως να εκμεταλλευτούμε και το γεγονός ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια στην τελική ευθεία, δεν έχουν κλείσει οι διαπραγματεύσεις. Βλέπετε ότι έχουμε κάπως προσαρμοστεί στην κατάσταση πραγμάτων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό που θα δείτε θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε ως σημείο εκκίνησης. Μας ενδιαφέρει να σεβαστούμε τις καταληκτικές ημερομηνίες της ε, συνθήκης. Προτού πάντως συνέλθει η Επιτροπή Συνδιαλλαγής, έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε αυτά τα οποία αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο στο φως των διαπραγματεύσεων για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές. Και φυσικά μπορούμε να τροποποιήσουμε τη διορθωτική επιστολή σε σχέση με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Έρχομαι στην επόμενη διαφάνεια τώρα. Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών. Οι πιστώσεις υποχρεώσεων ακολουθούν την κατανομή που είχε παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής σας στις 27 Μαρτίου. Υπάρχει όμως μια μεγάλη τροποποίηση υπάρχει μια εμπροστοφόρτιση των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ανεργίας των νέων για το 2014-2015. Αυτή είναι η βασική τροποποίηση του προφίλ των προτάσεων της 27ης Μαρτίου. Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, βασίζονται σε ένα πλήρη προϋπολογισμό για το 2014, αλλά είναι κάτω από την οροφή του 2013. Εκμεταλλευόμαστε όμως ό,τι περιθώριο έχουμε μέχρι την οροφή για τις πληρωμές. Λέμε λοιπόν ότι οι πληρωμές του 2014 δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν την οροφή αυτή. Και φυσικά όταν φτάσουμε στην τελική συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου μπορούμε να έχουμε μια διορθωτική επιστολή. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες. Αναφέρονται ήδη ως γνωστόν ότι δίνουμε αυτή την ιδιαίτερη εμποστοφόρτιση για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων. Έχουμε μία πρόβλεψη σε ό,τι αφορά την παροχή ρευστότητος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και αυτή πολύ σημαντική, αλλά πάνω απ' όλα ο προϋπολογισμός του 2014 θα πρέπει να είναι ένα επενδυτικό εργαλείο. Επομένως, η εστίασή του είναι στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να λοιπόν ένα εργαλείο επενδύσεων για τις περιφέρειες της Ευρώπης και τους άλλους ωφελούμενους και δικαιούχους του προϋπολογισμού. Είναι μέσα στη φύση του προϋπολογισμού όμως ότι ο προϋπολογισμός του 2014, εφόσον είμαστε στην αρχή μιας περίοδου σχεδιασμού, είναι ένας γεφυρωτικού χαρακτήρα προϋπολογισμός με όλες αυτές τις παράλληλες μορφές περιορισμού για τα θέματα διοικητικών δαπανών. Βρισκόμαστε λοιπόν στην αρχή της μείωσης θέσεων στην δίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε από το 2013 και αυτό θα συνεχίσει για το επόμενο διάστημα 5 ετών. Η επόμενη τώρα διαφάνεια Βλέπετε πόσο ενδιαφέρουσα είναι η δομή των πληρωμών που είναι, όπως υπογράμμισα και πριν, ο πρώτος χρόνος των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020. Για πολλά σχέδια θα υπάρξει φυσικά αργή εκκίνηση για την εκταμίευση και φυσικά έχουμε την εμπειρία του παρελθόντος. Η νέα όμως νομική βάση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, ώστε οι προτάσεις για σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Έχουμε δώσει λοιπόν ιδιαίτερη εστίαση στις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων που έχουν, όπως είπα, σαν εστίαση ανταγωνιστικότητα, θέσεις απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη. Κάτι που είναι επίσης σημαντικό να ξέρει κανείς είναι ότι το χάσμα μεταξύ πληρωμών και υποχρεώσεων έχει τέτοια μορφή ώστε να μην ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των λεγόμενων ραλ, των υπολείπων προς εκταμίευση, γιατί στο παρελθόν αυτό το χάσμα είχε φτάσει μέχρι και 18 δισεκατομμύρια. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε αυτό το ρυθμό αυξήσεως των ραλ και αυτό φυσικά θα διορθωθεί και με τον διορθωτικό προϋπολογισμό του 2013. Βλέπετε τώρα τη δομή των πληρωμών που είναι, όπως είπα, η γέφυρα μεταξύ του παλιού και του καινούριου. 14% είναι ε, για την ε, διοίκηση και την γεωργία. Αυτά είναι τα ίδια σε επίπεδο πληρωμών και υποχρεώσεων. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι υπάρχουσες υποχρεώσεις, δηλαδή 70% του, πληρωμού, του, προϋπολογισμού πληρωμών, καλύπτουν 70,7 δισεκατομμύρια. 70,7 δισεκατομμύρια λοιπόν οι πιστώσεις αυτές που, που αντιπροσωπεύουν το 52% του προϋπολογισμού. Ο γεφυρωτικός χαρακτήρας είναι να κλείσουν τα προηγούμενα προγράμματα χωρίς νέες υποχρεώσεις και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο του προϋπολογισμού 2014 να καλύψουμε τις ήδη συναυτήσεις υποχρεώσεις και θα είμαστε έτσι έτοιμοι να μειώσουμε κατά το 1 τρίτο όπως είπα προηγουμένως τα ράλ τα οποία υπάρχουν μέχρι το τέλος των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. γιατί στο τέλος του, 2000, του 2013 θα ήταν 200 ε, δισεκατομμύρια τα ΡΑΛ και αφού καταβάλουμε περίπου 70 δισεκατομμύρια θα μειωθούν κατά ένα τρίτο. Στο τέλος του πίνακα αυτού βλέπετε πόσο μικρές είναι οι υποχρεώσεις που αφορούν σύναψη υποχρεώσεων για νέα προγράμματα. Χρειάζεται φυσικά να γίνουν προπαρασκευαστικές εργασίες, αλλά αυτά καλύπτουν μόνο 10 δισεκατομμύρια και πρόκειται για προχρηματοδότηση ορισμένων σχεδίων και έτσι διατηρούμε το όριο του 1% του Εισοδήματο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξεπερνάμε αυτό το όριο. Αυτό λοιπόν για τις πληρωμές. Έχετε ένα πίνακα στη συνέχεια που βλέπετε τις ε, κατηγορίες του προϋπολογισμού. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στο κατάλληλο πλαίσιο. Και αυτό θέλω να τονίσω, το 2014 δεν είναι ένα έτος γέφυρα, αλλά είναι ένα έτος το πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της εξέλιξης μεταξύ 2014 και 2020. Όπως είπαμε, η εστίαση είναι περισσότερο στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα. Και βλέπετε και μόνοι σας πόσο αυξάνονται αυτές οι, οι, αυτά τα κονδύλια. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή σε αυτά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Δεν περιλαμβάνονται στις δημοσιονομικές προοπτικές. Έχουμε δύο κατηγορίες που είναι εκτός και αυτό γίνεται θεληματικά. Είναι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, αντιμετωπίσεις των προβλημάτων της ε, παγκοσμιοποίησης και το, το αποθεματικό για την έκτακτη βοήθεια. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να σεβαστούμε την αρχή της κινητοποίησης αυτών των εργαλείων γιατί το κοινωνικό ταμείο, το ταμείο ευελιξίας και το ταμείο αλληλεγγύης έχουν διαφορετική μορφή. Εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις αρχές των ε, πληρωμών και των υποχρεώσεων για τα θέματα αυτά που, είναι, που ξεπερνούν βέβαια την οροφή και γι' αυτό είναι εκτός των δημοσιονομικών προοπτικών. Τώρα βλέπετε μια εικόνα που είναι πιο συνολική συγκρίνοντας επταετής δημοσιονομικές προοπτικές. Βλέπετε ότι το ότι ξεκινάμε με αργό ρυθμό αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ευκαιριών επένδυσης που μπορούμε να δώσουμε στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν μπορούμε να εστιάσουμε περισσότερο στα σημαντικά θέματα. για τις ε, ευκαιρίες που λείπουν σε σχέση με τις επενδύσεις. Προφανώς η, το, η διευκόλυνση Connecting Europe είναι σχετικά καινούριο στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει το χαρακτήρα ενός προγράμματος ανάκαμψης και μπορούμε μονάχα να το συγκρίνουμε με κάτι το οποίο δεν έφερε το όνομα του Connecting Europe. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα για το μέλλον. Υπάρχουν βέβαια κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με ενεργειακά θέματα για όλα αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση έστω μερική. Και βλέπετε εδώ πέρα κάποιες διαφάνειες που δείχνουν την ε, εξέλιξη των δαπανών που βρίσκονται στο πλαίσιο της ε, ανταγωνιστικότητος, της συνοχής, της ε, εφηβούς και περιεκτικής ανάπτυξης κτλ. και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα δεν περιλαμβάνεται η, ο προϋπολογισμός ο Για τα θέματα συνοχής βλέπετε την επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε και τη φύση των σχεδίων που έχουν να κάνουν με τη συνοχή. Δεν με φοβίζει αυτή η πτώση που βλέπετε το 2014. Είναι απόλυτα φυσιολογική. Το θέμα είναι να έχουμε αρκετή χρηματοδότηση στο τέλος όταν τα προγράμματα έχουν οριμάσει. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα ράλ τα οποία έχουν δημιουργηθεί τη στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Δηλαδή μέσα στο 2014 2015 να καλύψουμε τις ήδη συναυτήσεις υποχρεώσεις γιατί αυτό είναι απαραίτητο για την ισορροπία των οικονομικών της Ευρώπης. Και μετά θα ξεκινήσουμε με νέα χρήματα για τα επόμενα πρόγραμματα, όχι μονάχα, που ξεκινάνε όχι μονάχα με μικρή ε, προχρηματοδότηση, αλλά και με ενδιάμεσες πληρωμές για το μέλλον. Και αυτό φυσικά θα αντανακλάται στις ε, πιστός υποχρεώσεων. Η τελευταία διαφάνεια περιλαμβάνει και τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Πάλι υπάρχει ε, ένα χαμηλό σημείο το 2014, αλλά αυτό οφείλεται ότι ξεκινάμε μια νέα γενιά προγραμμάτων. Και στη συνέχεια έχουμε την κατανομή σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα προγράμματα ναυαρχίδος. Έχουμε την πρωτοβουλία Ευρώπη 2020, έχουμε τις πρωτοβουλίες Ναυαρχίδος. τις εμβληματικές ε, αυτές πρωτοβουλίες και εδώ βλέπετε τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση στην ψηφιακή αζέντα για την Ευρώπη, για τις νέες ε, δεξιότητες, τη βιομηχανική πολιτική. Με τον τρόπο αυτό ο προϋπολογισμός αυτός μπορεί να ενισχύσει τις λεγόμενες εμβληματικές πρωτοβουλίες για το 2020. Έρχομαι στο επόμενο σημείο που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο θα συζητηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή όχι στα περιθώρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νομίζω και έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη. Είναι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ήταν και δική σας πρόταση βέβαια να υπάρξει αυτή η εμπροστοφόρτιση στο βαθμό του δυνατού. Χρησιμοποιούμε λοιπόν όλα αυτά που μπορούν να μπουν στην πρωτοβουλία για τους νέους και έχουμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια, το 2014 και 2015. Και φυσικά εδώ συμβάλλει και το Ταμείο Συνοχής. Έτσι έχουμε μια επανακατανομή των υποοροφών στις ε, κατηγορίες 1α και 1β. Παίρνουμε λεφτά από κάποια προγράμματα τα οποία αναμένουμε ότι θα αργήσουν να προχωρήσουν προγράμματα ενέργειας παραδείγματο χάρη στο Connecting Europe, εδαφική συνοχή η οποία ακόμα δεν έχει τύχει συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων και επομένως θα, θα καθυστερήσει η έναρξή της και το, τη συνοχή στην Ευρώπη μέσα στο Connecting Europe. Μετά από αυτά μπορούμε να εμπροστοφορτήσουμε τις υποχρεώσεις για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην απασχόληση των νέων για αυτούς που είναι σε ηλικία 15 έως 24 χρονών σε περιοχές όπου ξεπερνάει η ανεργία των νέων το 25%. Αν δείτε λοιπόν αυτό το πίνακα σε σχέση με την εμπροστοφόρτιση, Βλέπετε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς επαρκή χρηματοδότηση για το, επο, για το υπόλοιπο κομμάτι της ε, δημοσιονομικής περίοδου. 2014 με 15 είναι μονάχα η Αλλά το κοινωνικό ταμείο έχει πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση, η οποία θα πρέπει να φτάσει περίπου τα 80 δισεκατομμύρια. Ξέρω ότι υπάρχει και κάποια διαμάχη για το ποιο θα πρέπει να είναι το συνολικό όριο του κοινωνικού ταμείου μέσα στα διαρθρωτικά ταμεία. Αλλά πρέπει ένα μεγάλο μέρος αυτών των κονδυλίων να χρησιμοποιηθούν για να δώσουμε μια εγγύηση προς τους νέους για την απασχόληση και έτσι μπορούμε να κάνουμε λειτουργική αυτή την εγγύηση για τους νέους. Δεν είναι λειτουργικό γενικά παρά μόνο σε δύο-τρεις χώρες. Απαιτείται λοιπόν να κινητοποιήσουμε στοχευμένες μορφές χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη περίπτωση για να καλύψουμε την ανεργία των νέων, όπως επίσης και χρήματα από το κοινωνικό ταμείο για να μπορέσουμε να καλύψουμε την υπόλοιπη περίοδο. Για την υπόλοιπη λοιπόν περίοδο που είχαμε μηδέν για την, για την ανεργία των νέων επειδή έχει γίνει έμπροσθεν φόρτιση θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά ότι το κοινωνικό ταμείο θα μπορέσει να προσφέρει και να χρησιμοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή για το στόχο αυτό. Τώρα, επίσης ε, επίγον θέμα είναι το πώς ε, θα προχωρήσουμε στην ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει επαρκής ρευστότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε μέσα, πραγματικά μέσα, όχι μόνο πολιτικές ανακοινώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε ε, έσοδα από το Horizon 2020, από τα διαρθρωτικά ταμεία, από το Ταμείο Συνοχής, ε, να συνδυάσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε να λειτουργήσουν σαν μοχλός για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων. Έχετε μπροστά σας τα προγράμματα τα οποία μπορεί να συνδυαστούν. Και υπάρχει και το θέμα της εθελοντικής συμμετοχής και των Ευρωπαϊκών Διαφορετικών Ταμείων και των Επενδυτικών ε, ταμείων και μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως όλα αυτά μπορεί να μην είναι υψηλά ποσά, αλλά μπορούν να ε, μοχλεύσουν την έβρεση χρημάτων από τον ιδιωτικό τομέα και να καλύψουμε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον τρόπο αυτό. Ε, είναι κάτι το οποίο ε, αν δεν υπάρξει βέβαια συμφωνία ε, για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές ε, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα το οποίο δείχνει ότι δυνατότητες βελτίωσης της ρευστότητας των μικρομεσαίων υπάρχουν. Και τώρα περνάω σε ένα τμήμα θα έλεγα της παρουσίασης τίτλο, ανατίτλο δεν θα ασχολιάσω πάρα πολύ σε επίπεδο λεπτομέρειας. Όσο θα περάσει ο χρόνος, τόσο σε μεγαλύτερο βάθος θα περάσουμε σε όλους αυτούς τους τομείς. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να διαφοροποιήσουμε στο 2014 το τι μπορεί να φορτωθεί αμέσως, τι είναι όμως αυτό το οποίο ξεκινάει και απαιτεί ιδιαίτερα έντονες ικανότητες διαχείρισης και από πλευράς των κρατών μελών. Απαιτείται μια επίδειξη διαχειριστικής δυνότητας από πλευράς των κρατών μελών, το Horizon, το Horizon σαν παράδειγμα. Να είμαι ειλικρινής, εγώ νομίζω ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες για έμπροσθεν φόρτιση, και νομίζω ότι με αυτό συμφωνείτε και εσείς στα πλαίσια αυτών που ακούω για τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές ε, πλαίσιο. Υπάρχει δυνατότητα για τέτοιου είδους προγράμματα να υπάρξει ένα τμήμα, ένα ποσοστό ε, εμπροστοφόρτωσης. Αλλά το Horizon αφορά συγκεκριμένα προγράμματα, είναι κάτι το οποίο ξεκινά με αργή ταχύτητα και καλείται να επιταχυνθεί ε, σε ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν αυτήν την ευρύτερη εικόνα της εξέλιξης της κατάστασης ε, στο 1α για το Horizon 2020. Τώρα, το Ταμείο Connecting Europe δεν είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Απλά εξακολουθούμε εμείς να συλλέγουμε κάποια στοιχεία διαμεθοριακών συνδέσεων να τα σωρεύσουμε και να τα συγκρίνουμε με το Connecting Europe. Ε, το Erasmus ε, νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη για τον επόμενο ε, δημοσιονομικό ορίζοντα. Στο δεύτερο τμήμα του 1α μιλάμε για τη συνοχή και εδώ πρέπει να το μελετήσουμε προσεκτικά, απλά να επιστήσω την προσοχή σας Ο Ιβάιλο τα ξέρει καλύτερα, ο Ράιμερ επίσης. Δεν θα σχολιάσω όμως τίποτα σε σχέση με αυτό το, σε αυτή τη φάση, τα πράγματα είναι ακόμα ανοιχτά. Πάντως κάποιες πιστώσεις ήδη είναι στο προϋπολογισμό άνω των 360 εκατομμυρίων ευρώ αλλά ακολουθούν μάλλον πολλά ερωτηματικά για το πώς θα, σε πού θα καταλήξουμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Τώρα στον τίτλο 2. Θα έλεγα ο τίτλος 2 είναι ο πιο σταθερός από όλους. Αυτό είναι άλλωστε και η λογική των διαπραγματεύσεων. Όταν κάτι βγαίνει από τη μόδα τότε ξεκινούν οι πραγματικές διαπραγματεύσεις και αυτό φαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση για το 14. Στους άλλους τομείς είχαμε προγράμματα τα οποία ξεκινούν με χαμηλή ταχύτητα και επιταχύνων σαν αυτοκίνητα με μηχανές πετρελαίου. Ενώ τώρα έχουμε προγράμματα τα οποία ξεκινούν κανονικά, με μια τακτική θα έλεγα ε, ταχύτητα και δεν μας απασχολεί ε, η διαφορά ε, στην έναρξη του προγράμματος, εφαρμογής του προγράμματος. Έχουμε επίσης και το LIFE, ένα συγκεκριμένο ε, πρόγραμμα στο οποίο έχουν υπάρξει αρκετές υποσχέσεις και αυτό το λέω για την Όλγα. Το LIFE είναι ένα τμήμα μόνο του τι είναι διαθέσιμο μέσα από το mainstreaming. και υπάρχει ανάγκη εδώ για χρήση και χρημάτων από τα Ταμεία Συνοχής για την επεξεργασία των αποβλήτων, για τον καθαρισμό των υδάτων κτλ. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες χρήσης των πιστώσεων για, την, ε, για τον καθαρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, το επόμενο είναι η ιδιότητα του πολίτη και θέματα ασφάλειας. Να επιστήσω την προσοχή σας εδώ στο τι σημαίνει ε, η λειτουργία κάποιων ταμείων όπως για τη μετανάστευση κτλ. Αυτά δεν είναι βέβαια περιστρεφόμενα ταμεία. Έχουμε να κάνουμε με το αυτό που ονομάζουμε sharp management. Περιμένουμε τα προγράμματα από τα κράτη-μέλη και μετά θα δώσουμε τα χρήματα. Σίγουρα και εδώ ξεκινάμε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, συνειδητοποιούμε όμως ότι τα θέματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη και το τι συμβαίνει στη Συρία. Η Συρία προς το παρόν μας απασχολεί μόνο μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας το 2014. κάτω από τις ισχύουσες σήμερα συνθήκες. Πάντως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι θα ακολουθήσει αυτή την πολύ σοβαρή κατάσταση της σύγκρουσης στη Συρία. Τώρα για την ανάπτυξη. Αυτοί που ξεκινούν αργά, ναι μεν ξεκινούν αργά, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε επαρκή χρηματοδότηση. Τώρα για το Creative Europe, ε, Δημιουργική Ευρώπη τμήμα του Media. Εδώ τίθεται το θέμα της exception culturelle, λέει στα γαλλικά και ο και πολιτιστική εξαίρεση. Αυτό αφορά και το πρόγραμμα Media. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα εδώ και στα πλαίσια ε, του Creative Europe. Τώρα περνάμε στο Global Europe. Αυτό το οποίο θα πρέπει να φορτωθεί άμεσα είναι το κομμάτι που καλύπτει την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό το οποίο μειούται είναι η προενταξιακή βοήθεια. Και αυτό γιατί η Κροατία περνάει στην επόμενη κατηγορία, θα γίνει πλήρες μέλος. Ως εκ τούτου λοιπόν θα μάλιστα ακούσαμε και κάποια θετικά για τον διορθωτικό προϋπολογισμό, τον μικρό που αφορά την Κροατία σήμερα το πρωί. Το 2013 υπήρξε ισχυρή φόρτωση στον τομέα αυτό, γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν θα τα ξεπεράσουμε τα επίπεδα αυτά το 2014. Στον τίτλο 4 τα πράγματα είναι αρκετά καλά πάντως, να μην ξεχνάτε ότι στο μέλλον έχουμε επίσης και το αποθεματικό για την κατεπίγουσα βοήθεια εκτός ορίων τώρα. Το επόμενο ευαίσθητο θέμα είναι το θέμα της διοίκησης του διοικητικού προϋπολογισμού. Θα ήθελα εξ αρχής να σας ε, δείξω την, το μεσαίο αν θέλετε σχήμα. Βλέπετε εδώ κάποια σταθερά ποσοστά. 39% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Συνολικής Δαπάνης, τα υπόλοιπα όργανα 42% μαζί με το Κοινοβούλιο, και το 19% το κοινό είναι το πρόβλημα. Ακόμα και με τους μεγαλύτερους δυνατούς περιορισμούς στην διοίκηση, που αυτός είναι ξεκάθαρα το λέω στόχος μας, ε, και εδώ δεν συμπεριλαμβάνουμε την Κροατία, Αυτό το οποίο είναι σαφές εδώ είναι οι συντάξεις. Οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 6% το 2014. 7% όχι 6% το 14%. Όποιες και να είναι οι προσπάθειές μας και γίνονται και κάποιες εξοικονομήσεις και στα σχολεία, το ύψος της κατηγορίας αυτής, οι πιστώσεις που, απαιτεί, η κατηγορία αυτή είναι ε, μεγάλες. Λοιπόν, περιορισμός το διοικητικό κόστος, αύξηση του συνταξιοδοτικού κόστους και το ένα με το άλλο δυστυχώς δεν, το ένα μάλλον δεν καλύπτει το άλλο. Οι αυξήσει λοιπόν αυξάνονται. Τα έξοδα για τα άλλα όργανα παρά τη διεύρυνση προς την Κροατία, αν συγκρίνουμε τα 14 με το 12 θα δούμε ότι δεν έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση. Λοιπόν, οι δαπάνες τώρα για τη διοίκηση, όπως είπα, λαμβάνουμε υπόψη την πιθανότητα να παγώσουν οι μισθοί το 13 και το 14. Υπάρχουν κάποιες μικρές μειώσεις. Έτσι κι αλλιώ εσεί εμπλέκεστε σε αυτή τη διαδικασία και θα αξιολογήσετε τον πίνακα που σας παρουσιάζω. Ο επόμενος πίνακας αφορά τις θέσεις, όχι δαπάνες, όχι πιστώσεις, όχι χρήματα, αλλά προσωπικό, θέσεις προσωπικού. Εμείς προχωράμε σταδιακά στη μείωση του προσωπικού κατά 1% κατέτος, ξεκινήσαμε το 2013. Ακολουθούν όλα τα όργανα αυτή τη λογική, δεν είναι εύκολο, εφόσον έχουμε ταυτόχρονα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση νέες αρμοδιότητες. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι τα καταφέρνουμε εδώ και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τις προσπάθειες τις οποίες κάναμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει εμείς να καλύψουμε με 200 θέσεις την τελευταία φέτα θέσεων για την Κροατία. Παρόλα αυτά μειώνουμε τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων μας στο οργανόγραμμά μας για το 2014. Αυτή δεν είναι η πλήρης βέβαια εικόνα των διοικητικών δαπανών γιατί έχουμε και κάποια στοιχεία των διοικητικών δαπανών που βρίσκονται εκτός του τίτλου 5. Επαναλαμβάνω ότι πράγματι και με ικανοποίηση το λέω αυτό, ότι υπάρχουν ε, περιοριστικές τάσεις και στον τίτλο 5 και για τα εξωτερικά γραφεία και για το προσωρινό προσωπικό και για ό,τι βρίσκεται εκτός των τακτών διοικητικών δαπανών. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις, οι προβλέψεις που κάνουμε, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αριθμητικές προτάσεις. Είναι και θέματα αρχών που τίθενται εδώ. Έχουμε απλοποιήσει την ονοματολογία, έχουμε περάσει ορισμένα προγράμματα μέσω της διαδικασίας mainstreaming και για τις δηλώσεις των προγραμμάτων οι αριθμοί που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αντικαθιστούν τις δηλώσεις δραστηριότητας που είχαμε προηγουμένως. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα της γέφυρας ανάμεσα στον παλιό προϋπολογισμό και τον καινούριο. Αυτές είναι οι προβλέψεις για το 2014. Δεν σας κίνησα, έχετε ανοιχτά μάτια ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, όχι μόνο δεν κοιμήσατε το ακροατήριο, αλλά σίγουρα εκτίμησε και ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερος για τα λεγόμενά σας. Να δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στον εισηγητή κύριο Γένσεν και να πω ότι δυστυχώς ε, δεν θα μπορέσει να κάτσει για πολλή ώρα στη δική μας συνεδρίαση, έχει άλλες υποχρεώσεις. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι διαφωνεί ε, με αυτά που είπατε. Η κυρία Γένσεν λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως έχω μεγαλύτερο λόγο από ότι άλλοι ε, για αυτό το προπολογισμό. Σημείο κίνηση είναι το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, για το οποίο δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία. Εκτιλήσονται οι διαπραγματεύσει και βλέπω ότι το περίγραμμα που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση του προϋπολογισμού της ε, είναι ένα περίγραμμα το οποίο βασίζεται στη Συμφωνία Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Φεβρουαρίου. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο και είναι κατά τη διαφορετικό από την ανάλυση του προϋπολογισμού έτσι όπως την είχαμε δει μέχρι σήμερα, διότι τώρα είναι έμπροσθεν η φόρτιση της πρωτοβουλίας για τους νέους. Σίγουρα θα δείτε τη στήριξη του Κοινοβουλίου στην πρόταση αυτή παρόλο που πρέπει να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας στην πρωτοβουλία για τους νέους και μετά το 2015 να μην χρησιμοποιούνται μόνο τα κοινωνικά κονδύλια, το κοινωνικό ταμείο και το καθεξής. Βλέπω ότι προσπαθείτε να αποκαταστήσετε κάπως τη ζημιά που έχει γίνει στο Horizon 2020. Και αυτό είναι ανησυχία δικιά μας πράγματι. Το Συμβούλιο προσπάθησε τα μάλα να μας πείσει ότι πολύ περισσότερα κονδύλια θα δοθούν στην έρευνα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ωστόσο, δεν έχουμε καθόλου αύξηση για φέτος και πολύ βραδία αύξηση των κονδυλίων για το σύνολο της ε, περίοδου, της προγραμματικής. Και λέτε ότι ξεκινούμε με πτώση. Θα το δούμε αυτό σε συνεργασία με την Επιτροπή Ήτρε και θα δούμε ποια προγράμματα θα πληγούν περισσότερο, διότι το Horizon 2020 καλύπτει πολλά και διαφορετικά προγράμματα. Προγράμματα ανταλλαγών, για παράδειγμα, τα οποία κάλλιστα μπορούν να συνεχιστούν ε, και μπορούν να υλοποιηθούν ε, και μάλιστα πολύ γρήγορα. Το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής και δεν άκουσα καμία απάντηση ως προς αυτό. Η γεφύρωση για αυτή τη χρονιά. Έχουμε εκρεμεί το σχέδιο, το, το σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού για το 2012 τα δύο δις που κλήθηκαν τα κράτη να πληρώσουν. εκρεμίσει δηλαδή λογαριασμοί από αυτή τη χρονιά στην επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και αν δεν έχουμε το σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού υπαριθμών 2, τα υπολείποντα 3,9 δις που, για τα οποία δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο, πώς θα είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εσείς λέτε ότι πρακτικά δεν υπάρχουν περιθώρια. Και από εκεί και πέρα. Εκτός από την αναφορά στην έρευνα και στην πρωτοβουλία για τους νέους, αναφερθήκατε και στο Global Europe. Και η πολιτική εξωτερικών υποθέσεων ξέρετε ότι ήταν κάπως περίεργη ε, σε θέματα προϋπολογισμού θα είναι πρόβλημα, το οποίο θα αποκτήσετε σίγουρα με μας. Θα έχετε με μας πρόβλημα ως προς αυτό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Του χρόνου θα μειωθεί κατά 12% η δαπάνη για το Global Europe. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο δεδομένης της κατάστασης στη Συρία. Αυτή η μείωση του 12% πώς μπορούμε να την εξηγήσουμε δεδομένης της κατάστασης των προσφύγων στα Παλαιστινιακά εδάφη και από αυτά. Πώς είναι εφικτό ε, κάτι τέτοιο με αυτή τη μείωση. Έχουμε κάποιες ε, μειώσεις στο cargo free, αλλά είναι σχεδόν 10% σε σχέση με το 2013. Όλος αυτός λοιπόν είναι ένας ε, χώρος που πλήττεται ιδιαιτέρως, δυστυχώς. Και τέλος, ως προς τη διοίκηση. Είχαμε τους προβληματισμούς της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ως προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανησυχεί κατά πόσο η υπηρεσία αυτή θα μπορέσει να ε, λειτουργήσει με τις περικοπές που της έχουν επιβληθεί. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Προ το παρόν αυτού του προβληματισμού, ήθελα να καταθέσω. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο, Ευχαριστώ την κυρία εισηγήτρια. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Σας προτείνω να συνοψίσετε τις ερωτήσεις σας. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να προβείτε σε ε, γενικές δηλώσεις και σχόλια. Και αποφύγετε επίσης παρακαλώ να επαναλαμβάνετε ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί, ε, για να μπορέσει ο Επίτροπος να απαντήσει σε όλους. Συντονία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση αυτή. Βεβαίω είναι δύσκολο κανεί να εμφορείται από ενθουσιασμό με την παρουσίασή σα, διότι ούτω ή άλλω είναι δύσκολο να είναι κανεί ενθουσιώδη για το 2014 ούτω ή άλλω, διότι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι βέβαια καινούριο αυτό, το γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι καθήκον μα, αλλά και προνόμιο αν θέλετε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα είμαι όσο τον πιο σύντομη. Έχω ένα ερώτημα, Παύλα, σχόλιο μεθοδολογικής φύσης. Ποια υπόθεση επιλέξατε για να βασιστείτε για το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014 από πλευράς νομικής βάσης, δηλαδή ως προς τις πιστώσεις και τις δεσμεύσεις. Ξέρουμε από το παρελθόν ότι ε, ε, για το Life Plus ε, ο πρόεδρός μας ήταν ο πατέρας αυτού του προγράμματος. Δεν ξέρω αν ακούτε κύριε πρόεδρε, κύριε Λαμασούρ, γιατί σας κολακεύω αυτή τη στιγμή. Η δουλειά που έγινε εκεί είναι ένα μάθημα για εμάς όλους. Ποια υπόθεση εργασίας έχετε επιλέξει για νομική βάση, πρώτης πρώτου του 2014, πριν από αυτή την ημερομηνία, μετά από αυτήν. Πάρα πολλά επηρεάζουν την εκτέλεση ε, των πιστώσεων, την υλοποίησή τους δηλαδή. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε παρακαλώ. Επιπρόσθετα. Σίγουρα οι συνάδελφοι θα απαριθμίσουν τις επιφυλάξεις που έχουν για κάθε ένα από τα κεφάλαια του προϋπολογισμού. Δεν έχουμε αρκετά χρήματα για τις αποστολές μας, για τα σχέδιά μας, για αυτά τα οποία χρειάζεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ επινηρό να βλέπουμε τα νούμερα που μας παρουσιάζεται. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλω όμως να αναφερθώ σε κάτι που με αφορά εμένα προσωπικά, με ενδιαφέρει αλλά και με ανησυχεί και αναφέρομαι στην πολιτική συνοχής στη σελίδα 10 της παρουσίασής σας. Αυτή η πτώση των εκταμιεύσεων ε, για θέματα συνοχής, αυτή η μείωση και ρωτώ, ε, είναι κάτι που με ανησυχεί και με προβληματίζει. Αυτή η μείωση συνδέεται με την πρόβλεψη ε, βάση της οποίας θα γίνουν πολύ λίγες εκταμιεύσεις την πρώτη χρονιά και περιλαμβάνεται και τις επιπρόσθετες εκταμιεύσεις που έχουν δοθεί από τα κράτη-μέλη για αυτή τη χρονιά. Θα ήταν καλό να το γνωρίζουμε. Και τελευταία παρατηρήσή μου κάπως συναισθηματικής φύσεως ε, που συνδέεται και με τη διοίκηση. Με τρομάζει το γεγονός ότι το κόστος των συντάξεων εκτινάσεται σε αστρονομικά ύψη και οι δαπάνες για τα ευρωπαϊκά σχολεία μειώνονται ε, δραματικά. Δεν με αφορά προσωπικά γιατί το παιδί μου το πάω στο βελγικό σχολείο. Ωστόσο είναι θέμα φιλοσοφικό, ιδεολογικό αν θέλετε. Πού οδεύομαι όταν οι επενδύσεις διοχετεύονται στις συντάξεις και όχι στη νέα γενιά. Αλλά είναι κάτι που θα συζητήσουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, Ευχαριστούμε Σιδονία, η οποία σίγουρα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερο το μέλλον των νέων. Προσωπικώς δεν... Ε, ε, τρέφω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι γίνεται με τις συντάξεις. Ο Σαλβαδόρ Καρίγα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να κάνουμε λεπτομερές, ε, λεπτομερείς παρουσιάσεις γιατί μόλις λάβαμε το κείμενο αυτό. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι καλό ότι παρουσιάζεται σήμερα ο προϋπολογισμός διότι έχουμε μια γενικότερη άποψη και θεώρηση για το που θα οδηγηθεί η γενικότερη συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η οποία συμφωνία και θα είναι και η βάση για όλες τις δεσμεύσεις και τις πιστώσεις και τις ε, πληρωμές. Σε κάθε περίπτωση είναι το πρώτο έτος το 2014 του του δημοσιονομικού πλαισίου, είναι το πρώτο έτος προγραμματισμού και πιστεύω ότι ο Επίτροπος και οι υπηρεσίες του έλαβαν τη σωστή απόφαση. Δηλαδή να έχουν χαμηλές πιστώσεις για την πρώτη χρονιά, διότι η πρώτη χρονιά προγραμματισμού ξέρουμε από πάντα ότι ε, στην πρώτη χρονιά οι εκταμιεύσεις φτάνουν σε χαμηλά επίπεδα. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό ε, των πιστώσεων την πρώτη χρονιά. Δεν πιστεύετε ότι μάλιστα η βραδία εφαρμογή όλων αυτών το πρώτο χρόνο θα είναι ακόμα πιο βραδία από ό,τι προβλέπετε. Μήπως είστε υπερβολικά αισιόδοξο ε, στις προβλέψεις σας για το 2014 αφού είναι το πρώτο έτος. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο ή ερώτηση. Δεύτερο, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και κυρίως εν ώψη Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, δηλαδή το περιθώριο πιστώσεων πληρωμών 2014 και της οροφής είναι μηδενικό περιθώριο, 0,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σχεδόν τίποτα. Άρα θα έχουμε συνδιαλλαγή το Νοέμβριο υπό συνθήκες αρκετά διαφορετικές ε, συγκριτικά με τις άλλες οικονομικές χρήσεις. Και θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα τιμήσει την δέσμευση που έχει αναλάβει ε, για τον προϋπολογισμό των πληρωμών από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε ότι θα έχουμε κάποιες ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί η ζωή των τριών θεσμικών οργάνων από πλευράς προϋπολογισμού βάσει των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Και συμμερίζομαι το σχόλιο της Ιδονίας για τις συντάξεις. Ερωτώ κύριε Επίτροπε, είναι βιώσιμες οι συντάξεις με το τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια. Οι ευρωπαϊκές συντάξεις είναι ένα θέμα ουσίας που σίγουρα θα κληθούμε να αναλύσουμε και να συζητήσουμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Οι συντάξεις διαρκούν τόσο όσο ισχύει το προσδόκιμο ζωής πολύ συχνά οι συντάξει επιταχύνουν την εξέλιξη των γεγονότων. Ε, η Χάιντερ, Ισπανία, σοσιαλιστές τώρα αυτή τη φορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, διότι μας παρουσιάσατε το σχέδιο προϋπολογισμού. Ήσασταν πολύ σαφείς ε, στην παρουσίασή σας, η οποία ήταν ιδιαίτερα χρωματισμένη με ένα σωρό διαγράμματα και πίνακες. Ωστόσο, ε, η μείωση του 10 και του 12% που επαναλαμβάνεται δεν μας ε, ε, δημιουργεί όρεξη να μπούμε στις λεπτομέρειες. Ίσως θα χρειαστούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα τα διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, οι ερωτήσεις μου είναι το, οι εξής. Πρώτον, σε σύγκριση με το 2013, σε ποια νούμερα βασιστήκατε. Γιατί έχουμε πέντε ε, τροποποιημένους προϋπολογισμούς επιτάπητος για το 2013, ε, με κάποιες διαφορές. Δεύτερον, έχει σχέση με αυτό που είπε ο Σαλβαδόρ για το περιθώριο στις ε, εκταμιεύσεις και πληρωμές, το οποίο περιθώριο είναι σχεδόν μηδαμινό ή ανύπαρκτο έχετε προβλέψει τις πληρωμές έτσι δεδομένου του γεγονότος ότι πράγματι θα λυθούν τα του 2013 και θα ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός για το 2013 και δεν θα έχουμε έλλειμμα. Γιατί έχουμε ένα περιθώριο 11 εκατομμυρίων ευρώ για το 2013 και τώρα δεν έχουμε κανένα. Το έχετε δηλαδή διαμορφώσει αυτή την άποψη θεωρώντας ως δεδομένο ότι θα είναι ισοσκελισμένο το του 2013 είναι εξαιρετικά περίπλοκο χωρίς περιθώριο για το 2014 να επιληθεί όποιο πρόβλημα ε, μπορεί να προκύψει. Και τρίτον, ως προς την έμπροσθεν φόρτιση. Είναι κάπως δύσκολο να γίνει αυτό σε, με ορίζοντα το 2020. Έχουμε την πολιτική για την έρευνα και την ανάπτυξη που μπαίνει στην κατηγορία 1α. Εάν γίνεται όλο και περισσότερη έμπροστα φόρτιση χωρίς να αλλάζουν οι οροφές, σίγουρα θα αναγκαστούμε να περικόψουμε από κάποια προγράμματα, όπως με το Youth Guarantee. Σίγουρα πολλά προγράμματα χρειάζονται κονδύλια. Μπορείτε να μου πείτε όμως ποια είναι αυτά που δεν θα τη χρειάζονταν. Όλα τη χρειάζονται. Ε, όλα χρειάζονται βοήθεια. Εάν κάποια δεν χρειάζονται τόσο πολλά χρήματα, τότε γιατί τα έχετε προϋπολογίσει. Είναι κάπως περίεργη η τεκμηριωσή σας. Άλλο είναι να θέσουμε προτεραιότητες, να πούμε ότι το Youth Guarantee έχει προτεραιότητα έναντι άλλων πολιτικών, αλλά το να κόβει κανείς ε, κονδύλια από κάποια προγράμματα λέγοντας ότι δεν θα τα χρειαστούν, είναι κάπως περίεργη η τεκμηρίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άιντα. Ο Γιάν Μιλντερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο που μας παρουσίασε το προϋπολογισμό του 2014. Κοιτάζοντας το έγγραφό του και τις διαφάνειες, το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι ότι οι διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές έχουν προχωρήσει πολύ και πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι όμως το οποίο ίσως είναι απρόπτο. Αν δεν γίνει συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές, τι θα κάνουμε με αυτόν τον προπολογισμό. Πού θα βρούμε τη νομική βάση, πώς θα μπορέσουμε να δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα. Βλέπω ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι για παλιά προγράμματα και είναι λίγα χρήματα για νέα προγράμματα και υπάρχουν φαντάζομαι ακόμα ελλείψεις στις νομικές βάσεις για αυτά τα προγράμματα. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση με αυτά τα καινούργια προγράμματα. Μας είπατε ότι είναι θετικό το ότι υπάρχει μια συμφωνία για την Κροατία. Μα το Συμβούλιο τη δέχτηκε όπως την παρουσίαση η Κομισιόν ή έκανε αλλαγές και αν έκανε αλλαγές, τι αλλαγές. Και εγώ χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερα χρήματα για τους νέους για την αντιμετώπιση της ανεργίας. <clears throat> Είναι ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά από πού έρχονται αυτά τα χρήματα και ποιε είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν. Και ένα ακόμα σημείωμα ο διορθωτικός προϋπολογισμός υπαριθμών 2 που ανέφερε η κυρία Γένσεν. Φαντάζομαι ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι θα εγκριθεί αυτός ο προϋπολογισμός υπαριθμών 2 όπως έχει υποσχεθεί το Συμβούλιο και βασίζεται στην υπόσχεση αυτή. Η Έλγα Τρίπελ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Επίτροπό μας για την παρουσίαση αυτή. Το πρώτο ερώτημά μου είναι το εξή. Υπάρχουν λόγοι για εμπροστοφόρτιση σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τους νέους, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι είναι αυτό το οποίο οπισθοφορτίζεται για να αντισταθμίσει αυτά τα χρήματα. <clears throat> Και επίση κύριε Επίτροπε, στην παρουσίασή σας είπατε ότι θέλετε να δώσετε μεγαλύτερη ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπω τη σελίδα τώρα 15. Και εδώ τίθεται το πολιτικό θέμα των προτεραιοτήτων. Βλέπω 26% μείωση για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 2,5% για το ορίζον 2020, 13,5% σε υποχρεώσεων και 24% και για τον έρασμο υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές κατά 12,7%. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που εμείς ως Κοινοβούλιο θέλαμε να δούμε και δεν συνάδει με αυτά που είπατε στην αρχή, ότι θέλετε να έχετε περισσότερη ρευστότητα, περισσότερη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τουλάχιστον από αυτή τη σελίδα που σας ανέφερα υπάρχουν σαφείς μειώσεις στο τομέα αυτό και στη σελίδα 7 τώρα έρθω Αν συγκρίνω τα χρήματα για ανταγωνιστικότητα και θέσεις εργασίας τα μειώνεται κατά 9%. Αλλά για τις αγορές που έχουν να κάνουν με την αγορά αυξάνεται κατά 0,3% και στην αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την ε, αλληλεία που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και τις νέες αυτές οικονομικές δραστηριότητες μειώνονται τα κονδύλια κατά 10%. Πού είναι λοιπόν αυτή η ισορροπία που λέτε. Αυξάνονται οι άμεσες πληρωμές και η γεωργία στη γεωργία, αλλά μειώνονται τα κονδύλια για την ανταγωνιστικότητα. Για μένα αυτή δεν είναι η σωστή ισορροπία και δεν έχει καμία σχέση με αυτήν με την δημοσιοσχεσίτικη παρουσίαση που κάνετε στην αρχή. Και η τελευταία μου παρουσίαση, παρατήρηση, συγγνώμη. Αυτά τα οποία δεν θα πληρωθούν από τον ε, Νοέμβριο του 2013 και αν μεταφερθούν στο 2014 αυτές οι εκταμείευσεις αν δεν γίνουν, τι επίπτωση θα έχουν στον προϋπολογισμό του 2014. Ευχαριστώ Έλγα. Η Άλντα Σόσα. Ευχαριστώ Αλά. Ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο. Θα ήθελα ξεκινώντας να τονίσω ότι μας δυσαρεστεί πάρα πολύ η στάση της Κομισιόν γιατί συμπεριφέρεται η Κομισιόν αν με τον, με, το, με τον τρόπο που φέρεται είναι σαν να θεωρεί δεδομένη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουάριο και παραγνωρίζει απόλυτα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θέλω να εκφράσω την αντίθεση της ομάδας μου σε σχέση με τις διάφορες δηλώσεις που έγιναν δημόσιες και από την Κομισιόν και από την Ιρλανδική Προεδρία σε σχέση με τις πολιετής ε, δημοσιονομικές προοπτικές στη στιγμή που δεν υπήρχε ακόμα τελική συμφωνία. Αλλά ας σταθώ τώρα στην πρόταση αυτή. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία επισημάνθηκαν ήδη, αλλά πρέπει να πω ότι προφανώς αυτή η πρόταση προϋπολογισμού για το 2014 είναι μια πρόταση που περιέχει τη λιτότητα και που η ομάδα μου δεν μπορεί να τη δεχτεί με τη μορφή που έχει. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη ανάλυση, όχι βέβαια σε όλες τις θέσεις, αλλά θέλω να ρωτήσω Πώς μπορείτε να μιλάτε για αύξηση της ανταγωνιστικότητος όταν βλέπω να υπάρχουν μειώσεις στον ορίζοντα 2020, 24% μειώσεις στις πληρωμές. Δεν είναι ψίχουλα αυτά. 13% μείωση στον έρασμο, στο κόσμος, κόσμο, συγγνώμη, που υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάλι και εκεί μειώνονται τα κονδύλια. Ενώ το Connecting, European, Connecting Europe Facility ουσιαστικά είναι στο μεγαλύτερο μέρος εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επομένως, τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο δημοσίων επενδύσεων ουσιαστικά δεν είναι επαρκή. Έρχομαι τώρα στις πολιτικές συνοχής στο σύνολό τους, όπου υπάρχει σημαντική περικοπή. Σε ό,τι αφορά τις νέες δράσεις, 3,6 δισεκατομμύρια έχουμε για την πρωτοβουλία της απασχόλησης των νέων και 0,4 δισεκατομμύρια για τη βοήθεια προς τους πιο ενδεείς στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα αστείο. Είναι κατά κάποιο τρόπο να κλείνουμε τα μάτια μας και να θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν νέα προγράμματα αυτού του είδους. Αυτό είναι αστείο. Επίση για την αγροτική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική η περικοπή που γίνεται. Έχουμε περικοπές για τις, το Ταμείο Μετανάστευσης και για το Άσυλο, που οπωσδήποτε είναι απαραίτητη χρηματοδότηση εκεί. Περιορίζεται και η χρηματοδότηση για την Δημιουργική Ευρώπη, για το πρόγραμμα Media. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει καμιά σχέση με την ιδέα της πολιτιστικής εξαίρεσης. Για μένα λοιπόν η Κομισιόν ουσιαστικά εγκαταλείπει την πολιτιστική εξαίρεση και θέλει να εφαρμόσει πλήρως τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με τις ΗΠΑ όπου η ευρωπαϊκή κουλτούρα θα εξαλειφθεί απόλυτα και δεν θα υπάρξει καμιά υποστήριξη προς αυτήν. Νομίζω ότι αρκετά σας έχω πει για να καταδείξω την δυσαρέσκεια της ομάδας μας με αυτή την πρόταση θα ήλπιζα ότι πέραν όλων αυτών που έχουν γίνει στο παρελθόν, η Κομισιόν δεν θα έφτανε να παρουσιάσει μία πρόταση αυτού του είδους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος Ashworth. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αντίθετα με άλλους ομιλητές, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο και να τον συγχαρώ για την πραγματιστική και λογική του πρόταση. Εν γέννη κύριε Επίτροπε, εγώ χαίρομαι που δέχεστε τις, ε, τα, τα κονδύλια όπως αναφέρθηκαν το Φεβρουάριο του 2013 Εγώ θα ήθελα βέβαια να υπάρξουν πιο ριζοσπαστικές αλλαγές, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνετε κάποια βήματα θετικά. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε για τις επενδύσεις στον προπολογισμό γιατί είναι αυτό το οποίο λείπει στην Ευρώπη σήμερα. Ανταποκρίνεστε επίσης σε κάποια από τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφερθήκατε στην πρωτοβουλία για τους νέους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι θέματα στα οποία θα έπρεπε να είχαμε παρέμβει πριν από αρκετό καιρό, αλλά έστω και τώρα. Σχετικά με την πρωτοβουλία για τους νέους, πράγματι δέχομαι ότι η έμπροσθεν φόρτωση είναι κάτι το ρεαλιστικό. Από την άλλη μου δημιουργούνται κάποιες ανησυχίες για την ικανότητα απορρόφησης ε, σε μικρό χρονικό διάστημα των ποσών αυτών. Τι ε, δυνατότητες απορροφητικότητας έχουμε και ε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Και αν πράγματι αυτό θα πρέπει να κάνουμε και για να το λέτε το πιστεύετε, γιατί να μην χρειάζονται περισσότερη τρέχουσα στήριξη γιατί τέτοια προγράμματα, το είπατε κι εσείς, θέλουν πολύ χρόνο έτσι ώστε να αποδώσουν καρπούς, οπότε θέλουν και μία συνέχεια και μία χρονική διάρκεια. Λοιπόν, σας συγχαίρω για την γενική σας κατεύθυνση, σας συγχαίρω για την αυστηρότητα σε εισαγωγικά του προϋπολογισμού σας και θα στηρίξω την πρότασή σας. Κύριε Επίτροπε, είδαμε ότι πράγματι καταφέρατε ε, να συνδυάσετε κάποιους πολύ δύσκολους παράγοντες. Μία ερώτηση για τον προϋπολογισμό λοιπόν του 2014. Ξέρετε ότι δεν έχει κλείσει ουσιαστικά ο προϋπολογισμός του 2013. Λόγω ακριβώς αυτού της ανόητης στάσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ιδίου αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και πραγματικά αυτά τα οποία προβλέπετε για το προσωπικό και οι μειώσεις για το προσωπικό είναι ελάχιστες, είναι γελία ελάχιστες και θα έπρεπε ε, να καταγγείλουμε αυτό, αυτή τη συμφωνία σαν σκάνδαλο. Θα συμφωνήσετε λοιπόν μαζί μου ότι θα υπάρξουν ε, συνέπειες για τη στάση αυτή. Ευχαριστώ συνάδελφε. Και Εγώ θα ήθελα να εκφράσω μια ανησυχία την οποία έχω και να θέσω και ένα ερώτημα. Η ανησυχία μου αναφέρεται στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Μιλάτε για τις ηλικίε 15 με 24, αν έχω καταλάβει καλά. Αν κάποιος αναλύσει τις στατιστικές με κάποια λεπτομέρεια, σε κάποια προσοχή, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι βρίσκονται σε περίοδο κατάρτισης. Εξαρτάται λοιπόν ιδιαίτερα με τους νέους οι οποίοι βρίσκονται σε περίοδο κατάρτισης και σπουδών στα πανεπιστήμια. Οπότε αυτοί συμπεριλαμβάνονται γιατί πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται γιατί τα πράγματα χειροτερεύουν από τα 24 και μετά, γιατί η κατάρτιση επαγγελματική και οι πανεπιστημιακές που τερματίζονται στα 24 και από εκεί ξεκινάει το δράμα των ανθρώπων αυτών από τα 24 μέχρι 29 που δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα να εργαστούν ούτε και να σπουδάσουν. Αν λοιπόν μπορέσουμε να σταθμίσουμε κάπως τα πράγματα έτσι ώστε να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι, δεν θα έχουμε πετύχει τον στόχο τον οποίο έχουμε ε, μπροστά μας, έχουμε θέσει. Σχετικά τώρα με τις διοικητικές δαπάνες, βλέπω ότι υπάρχει μια ουσιαστική μείωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά σχολεία, 5,7. Δεν ξέρω πώς δικαιολογείται αυτό το θέμα, γιατί ακριβώς εκεί Εκεί βλέπω να υπάρχουν οι πιο έντονες περικοπές στα ευρωπαϊκά σχολεία. Γιατί, ποια είναι η κατάσταση στα ευρωπαϊκά σχολεία, τι μας υποχρεώνει να έχουμε τόσο μεγάλη περικοπή για τα κονδυλία των ευρωπαϊκών σχολείων. Ευχαριστώ πολύ, Ιούτα Χάουγκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το γεγονός ότι ο Επίτροπος ήρθε πρώτα να μας παρουσιάσει εμάς τον προπολογισμό και μετά στην εμβρόντιτη κοινή γνώμη θα παρουσιάσει τον προπολογισμό μετά από εμά. Εγώ δεν είμαι βέβαια γενική εισηγήτρια για τα θέματα αυτά. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι σαφέ, ξέρουμε και το είπε και ο Επίτροπο, ακόμα και αν δεν μα αρέσει, ότι θα λειτουργήσει επί τη βάση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του, της 8ης Φεβρουαρίου. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα αυτής της στάσης της Κομισιόν. Έχω ένα ειδικό ερώτημα εδώ και να φέρω και τα ερωτήματα κάποιου αδέρφου. Το ειδικό αυτό ερώτημα είναι το εξής. Για το πρόγραμμα LIFE. Κατανοώ ότι το πρόγραμμα αυτό, το LIFE, ότι συνδέεται και με την Helga στο μυαλό του κυρίου Επιτρόπου με αυτά τα οποία υπήρχε έλεγα στην Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών. Αλλά είναι ενδιαφέρον το ότι και για τη συντόνια, για το απόγευμα, πιστεύετε ότι στον τελευταίο τρίλογο που θα γίνει με το Συμβούλιο ότι μπορούμε να κλείσουμε όλα αυτά τα θέματα εκτός από τα συγκεκριμένα αριθμητικά ποσά. τότε μπορούμε να προχωρήσουμε από την 1η Ιανουαρίου. Αλλά για τη χρηματοδότηση τώρα επανέρχομαι, η Κομισιόν. Στην πρότασή της για το πρόγραμμα LIFE είχε προτείνει 3,22 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Ακολούθησε η απόφαση του Συμβουλίου στις 8 Φεβρουαρίου και έχουμε μια ενδεικτική κατανομή κονδυλίων. Αυτή η ενδεικτική κατανομή κονδυλίων περιλαμβάνει και τα μικρότερα προγράμματα και το live που είχαν 3,057 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ στο έγγραφο που μας παρουσιάζεται και στη σελίδα 8 όπου πρόκειται για μερικά συγκεκριμένα προγράμματα και αναφέρεστε πάντα σε τιμές του 2011 Έχουμε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν δω τα στοιχεία για την εξέλιξη του προγράμματος LIFE, αν τα προσθέσω όλα αυτά, φτάνω στο 3,456 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι επίκριση αυτό. Τι ακριβώς είναι ρεαλιστικό και τι είναι πραγματικό. Πώς ακριβώς θα πρέπει να καταγράψω αυτό. Θα πάρει περισσότερα χρήματα το live από ό,τι στο παρελθόν. Δεν έχω καταλάβει. Δεν θέλω να σας επικρίνω, αλλά δεν μπορώ να αφήσω αυτό το θέμα χωρίς να το σχολιάσω και να πω τι ωραία, ναι, καλά και να μου πείτε στο τέλος, α, ήταν κάποιο τυπογραφικό λάθος και μόνο. Και τώρα το επόμενο σημείο. Εγώ θα ήθελα, όπως και ο Γιάνν Μίλντερ, τι ακριβώς θα γίνει αν στο ορατό μέλλον δεν υπάρξει πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι ακριβώς θα γίνει, τι θα γίνει με τη νομική βάση. Ξέρω ότι πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες νέες νομικές βάσεις, ενδεχομένως θα μπορέσει να γίνει αυτό. Αλλά το δεύτερο θέμα είναι και το ερώτημα που έθεσε ο πρόεδρος μας. Αν η ειδική συνεδρία που θα κάνουμε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Στρασβούργο βασιστεί στο ότι η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων έχει πάρει μια απόφαση αν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το οποίο αποφάσισε η Κορεπέρ και μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια με αυτό ή αν πρέπει να βασιστούμε σε κάτι άλλο. Τι ακριβώς ισχύει σε αυτήν την περίπτωση. Ευχαριστούμε Γιούτα. Σας απαντώ εγώ στο ερώτημά σας. Στην έκτακτη συνεδρίαση της Δευτέρας το βράδυ στο Στρασβούργο θα έχουμε στην ημερησία διάταξη ούτως ή άλλως με την επιφύλαξη της ε, συζήτησης στην Κορεπέρ σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να ψηφίσουμε τον ΤΑΠ 1. Θα έχουμε τον, τον, ε, διορθωτικό προϋπολογισμό 1, ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε για ένα κομμάτι του διορθωτικού 2, και θα πρέπει να σταθούμε και στις διαπραγματικές πολιτικές δημοσιονομικές πρόπτικες που θα έχουν λάβει μέρος, θα έχουν λάβει χώρα μάλλον, μέσα στα περιθώρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί με ποιο τρόπο αν καταλήξουν όλα αυτά σε πολιτική συμφωνία, θα μπορούσε μια έκτακτη σύνοδος της Κορεπέρ την ε, Παρασκευή να τα υλοποιήσει αυτά σε προτάσεις συγκεκριμένες πριν από τη δική μας συνεδρία στο Στρασβούργο τη Δευτέρα. Ούτως ή άλλως θα έχουμε μια ψηφοφορία για τον διορθωτικό προϋπολογισμό υποαριθμών 1. Ο Ντομινίκ Ρικέ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας παρουσίασε γιατί βασίζεται στα στοιχεία του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις πολιετήσεις δημοσιονομικές προοπτικές και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θα γίνει αν εφαρμοστεί αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα έχει ένα δρακόντιο χαρακτήρα. Κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πέραν της γενικής ε, διαδικασίας περικοπής σε επίπεδο ποσοστών. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση των πληρωμών τα πρώτα χρόνια για λόγους εκκίνησης ε, των προγραμμάτων. Αλλά αυτό σημαίνει ότι σε μια στιγμή που η Ευρώπη είναι σε ύφεση, που είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ενεργή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έτη 2013-2014 ουσιαστικά θα καταρρεύσει η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έτη αυτά, όχι μονάχα γιατί δεν θα έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα αυτά, αλλά και διότι θα μειωθεί και ο προϋπολογισμός για τα έτη αυτά. Αυτό καταδεικνύει λοιπόν με μεγάλη σαφήνεια τι ακριβώς θα γίνει. Παρά τις καμπύλες που ανεβαίνουν στη συνέχεια θα πρέπει να δει κανείς τα απόλυτα ποσά και την γούβας, στην οποία θα βρεθεί χρηματοδότηση το 2013-2014. Και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση λόγω της περικοπής των κονδυλίων στα ετήσια προγράμματα. Τώρα τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα, θέλω και εγώ όμως να θέσω ορισμένα. Το πρώτο ερώτημα, αν η πολιτική να εξαφανίζονται τα περιθώρια είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ευελιξίας. Το δεύτερο θέμα το πρόγραμμα για την ε, απασχόληση των νέων, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι. Δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε μια πολιτική πληρωμών η οποία να είναι εξαιρετικά στεναρή ακόμα και μέσα στην πολιτική λιτότητας. Αν το ξέραμε αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά σημαντικά πράγματα και σε άλλους τομείς. Όταν είναι τόσο δύσκολο λοιπόν να μπορέσουμε να καλύψουμε την έλλειψη προγραμμάτων, μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και σε άλλους τομείς αυτή τη διαδικασία. Για το ΑΑ τώρα, για το 1α μάλλον, έχουμε 12,5% για το Connecting Euro Europe Facility και υπάρχουν μεγάλα προγράμματα υποδομών για 16,2 ε, δισεκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς συνάδουν αυτά τα δύο. Επίσης η, η μείωση κατά 9,4% στο σημείο 3. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε μια τόσο μεγάλη μείωση όταν ε, υποδεχόμαστε και άλλο ένα κράτος ε, μέλος, αλλά και όταν υπάρχουν και οι εξελίξεις λόγω της προσθήκης του νέου κράτους μέλους στα θέματα του Σέγγεν. Αυτά είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θέσω στην Κομισιόν. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το έργο της Κομισιόν, αλλά εγώ ως εκπρόσωπος του ΕΛ θα σας πω και πιο λεπτομεριακά στοιχεία στην συνέχεια. Κύριος Γκοτμάνης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Είναι τα μέγιστα που μπορούσε να μας πει σήμερα και τα μέγιστα που μπορούσε να μας δώσει σήμερα. Θέλω να ε, ρωτήσω το εξής για την έμπροσθεν φόρτιση της ε, πρωτοβουλίας για τους νέους. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι ε, απότοκος του υπάρχοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Μέχρι τα τέλη αυτής της χρονιάς θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, δεν έχει επεκτάσεις. Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα. Πόσο καλά θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους του υφιστάμενου σχεδίου γιατί έτσι θα μπορούσαμε να κρίνουμε πόσο καλοί θα είμαστε όταν κληθούμε να υλοποιήσουμε την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Είναι σοβαρό το ερώτημα. Ε, στον τρίλογο, στον τριμερή διάλογο του οποίου είμαι μέλος, η Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, αλλά και άλλοι πετούν από το παράθυρο την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων λέγοντας ότι για αυτήν ε, τα χρήματα θα έρθουν από το κοινωνικό ταμείο και ούτω καθεξής. Όμως, η πρωτοβουλία για, τις για τους νέους είναι κοινωνικό πρόβλημα. Ποιος θα διαχειριστεί ε, το σχέδιο αυτό. Δεν θα λυθεί με την έμπροσθεν φόρτωση γιατί μπορεί να μην υπάρξουν σοβαρά αποτελέσματα. Και γιατί το φοβάμαι αυτό. Διότι ανάλυσα το ποσοστό των ε, κονδυλίων στο κοινωνικό ταμείο. Πόσα δίδονται άμεσα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σήμερα. Το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Είναι οι υπόλοιπε χώρες έτοιμες όταν η ανεργία των νέων ξεπερνά το 25% να υλοποιήσουν ταχύτατα την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη και τα τρία δις. Και ποιος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μεριμνήσει ότι ε, τα χρήματα αυτά δεν, δεν σπαταλώνται με πολύ πραγματικές εκφράσεις χωρίς πραγματικά να πιάνουν τόπο. 20 ε, Ιουνίου έχω τη δήλωση του Συμβουλίου, το έγγραφο το οποίο δόθηκε στα κρατη και έχουμε το άρθρο 9G, το συνολικό ε, περιθώριο των επιστώσεων για τους νέους και ούτε καθεξής. Τι κρύβεται δηλαδή εδώ από τις μη χρησιμοποιημένες, από τα μη χρησιμοποιημένα κονδύλια από άλλα άρθρα θα παρθούν τα χρήματα και θα έχουμε στην φόρτωση για το 2014. Δηλαδή τα μη χρησιμοποιηθέντα χρήματα και τίθεται και το ερώτημα θα υπάρξουν για να κάνουμε αυτή την περιβόητη έμπροσθεν φόρτωση, θα υπάρξουν κονδύλια χρησιμοποιητά. Αλλά και να υπάρξουν. Εγώ δεν είμαι κατά όλο αυτών. Ε, ερωτώ όμως τον Επίτροπο Είμαστε σοβαρά προετοιμασμένοι. Πόσα πολλά θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη και πώς θα καταφέρουμε να μην ε, δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα χωρίς να πιάσουν τόπο. Αυτά προς το παρόν, αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ πολύ. Εντίτ Εψόκ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχετε μια εξαιρετική ικανότητα δημιουργικής λογιστικής μας δείχνει ότι δεν βουλιάζει η βάρκα, ότι ανεβαίνει η οροφία, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, με τη δημιουργική αυτή διαχείριση ε, βουλοπλέουμε. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Για αυτό το κεφάλαιο, είστε έτοιμοι να πείτε όχι αν ανεβεί πάλι το κόστος είτε την επόμενη χρονιά και τις επόμενες. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια και χαίρομαι που είναι εδώ η Μόνικα Χολμάγερ και εκπλήσωμαι ότι κανείς δεν έχει θέσει ερώτημα ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω την αίσθηση, κύριε Επίτροπε, ότι δεσμεύεστε να μην υπάρξουν νέα μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μην υπάρξουν αλλαγές και πρέπει να απαριθμηθούν τα παλαιά μέλη. Δεν γίνεται καθόλου λόγος για την απαρίθμηση και η απαρίθμηση των μελών βάσει των τελευταίων εκλογών είναι στο 2,2% ενώ εσείς έχετε αναφέρει το ποσοστό του 1,7%. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτή τη διαφορά. Νομίζω ότι είναι κοινή αίσθηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει και η σύνταξη των μελών να μπει στο πρόγραμμα αυτό και να ευθυγραμμιστεί. Γιατί αυτό είναι και το μεγαλύτερο βάρος, ότι θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή ενιαία γραμμή για όλες τις συντάξεις. Όλα αυτά κάνουν την οικονομική χρήση σχεδόν αδύνατη στην εκτέλεσή της. Στη σελίδα 27 υπάρχει και ένα λάθος υπολογισμού η διαφορά δεν είναι 1,2% αλλά 2,4%. Έχετε βάλει και τα αριθμητικά στοιχεία για την Κροατία στη σελίδα 7. Δεν είναι 1,7 η διαφορά, αλλά 2,4. Στη σελίδα 27 λέει η μιλήτρια τώρα. Στη γραμμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο υπολογισμός είναι λάθος. αριθμητικά βασικό εκτός και αν έχετε προσθέσει κάτι για την Κροατία το οποίο δεν είναι εδώ. Η διαφορά δεν είναι 1,7 επαναλαμβάνω, είναι 2,4 στη σελίδα 27 ε, στην επικεφαλίδα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη γραμμή αυτή εν πάση Και τέλος, τα ευρωπαϊκά σχολεία θα συνεχίσουν να πηγαίνουν χέρι-χέρι με τι συντάξεις ή θα γίνουν μειώσεις και γίνονται μειώσεις στα ευρωπαϊκά σχολεία γιατί αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρωθεί για τις συντάξεις χωρίς να το μαθαίνει η κοινή γνώμη. Χαίρομαι ιδιαίτερος που η Συντονία το έθεσε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία αυτή για τους νέους σε ποια νομική βάση βασίζεται και σε ποιο βαθμό έχει διαμορφωθεί ήδη η νομική αυτή βάση ή θα υπάρξει κάποια άλλη βάση από τις πολυετής προοπτικές. Η Μόνικα Χολ, Χολμάιερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θέλω να διαμαρτυρηθώ έντονα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλειψε να ενημερώσει τους συζητητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι πρέπει να αλλάξουν τους αριθμούς, του, τους αριθμούς τους. Είμαστε η δεύτερη, το δεύτερο σκέλος της αρχής του προεπολισμού και περιμένουμε ότι η Κομισιόν τουλάχιστον θα έρθει σε επαφή με τον εισηγητή του Κοινοβουλίου και όταν θέλετε να έχετε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει εμείς να μπορούμε να προσαρμόσουμε τα ποσά βάσει του προϋπολογισμού. Υπάρχουν αλλαγές λοιπόν για τον κανονισμό των υπαλλήλων, αλλάζει επίσης το σύνολο του κόστους, δεν μας έχετε πληροφορήσει καθόλου για τα θέματα αυτά. Μίλησαμε με τον Επίτροπο πριν από δύο εβδομάδες για το κανόνα του 1% αλλά δεν μας είπε καθόλου η Κομισιόν ότι είναι έτοιμη να αλλάξει τα στοιχεία της χωρίς να ενημερώσει τον ε, εισηγητή του Κοινοβουλίου. Αντίθετα λέτε για τους υπαλλήλους της Κομισιόν, τους ε, υπάλληλους του Κοινοβουλίου κάτω από το επίπεδο του Διευθυντή και στη συνέχεια αφήνεται να διαρρεύσουν όλα αυτά τα στοιχεία από την Κομισιόν προς τους διαπραγματευτές, διαπραγματευτές χωρίς όμως αυτό να είναι επίσημη πρόταση. Μας τα δίνετε ανεπίσημα και δεν ξέρουμε τελικά τι είναι ουσιαστικό και τι είναι ανεπίσημο. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά παραγνωρίζετε και περιφρονείται τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα τηλέφωνο να είχατε σηκώσει θα μπορούσατε να έχετε επαφή μαζί μας. Θέλω να το πω αυτό, έχω ενοχληθεί πάρα πολύ και νομίζω και οι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται και θέλουν να συμβάλλουν στο να υπάρξει το κοινοβούλιο, να μπορέσει να υπάρξει προγραμματισμό από το κοινοβούλιο, δεν μπορούν να αποδεχτούν μια τέτοια στάση. Και αν έχουμε τα στοιχεία μόνο σήμερα, εγώ είδα ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουνε, μπορέσει να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν από εμά και δεν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ ημών για αυτά τα στοιχεία. Και για το 2013 εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα θέματα αυτά. Πρέπει να περιμένουμε την απόφαση για το, το θέμα αυτό. Δεύτερον, η Κομισιόν έχει αφαιρέσει 14,4 εκατομμύρια από αυτά τα οποία είχαμε ε, συμφωνήσει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, είπαμε ότι όταν έρθει ο νέος κανονισμός για τους υπαλλήλους θα έχουμε και το, την ανάγκη να προσαρμόσουμε όχι μόνο τον κανονισμό αλλά και τα κονδύλια. Η Κομισιόν θεώρησε ότι αυτό όμως μπορεί να το κάνει μόνη της χωρίς να ενημερώσει καθόλου το Κοινοβούλιο. Αλλά τα στοιχεία τώρα πια δεν ισχύουν, δεν ταιριάζουν αυτά τα στοιχεία που είχαμε εμεί στα χέρια μας με αυτά που λέει η Κομισιόν βγάλατε 14,4 εκατομμύρια, 0,7% από το 2014, 1,1% από το 2013. Με ποια βάση έχετε εσείς υπολογίσει αυτά τα ποσά πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό έχετε αφαιρέσει και τα κονδύλια για την Κροατία εδώ ή όχι. Γιατί εμείς είχαμε περιλάβει την Κροατία στους υπολογισμούς μας. Θα ήτανε πολύ καλό η Κομισιόν να μιλάει πρώτα με τους εισηγητές και μετά να κάνει τις τροποποιήσεις στα στοιχεία της. Θα ήταν κάτι πολύ εύκολο. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Άπειρες φορές έχουμε συζητήσει για τα θέματα αυτά, αλλά η Κομισιόν θεώρησε ότι δεν έχει καμία ανάγκη να έρθει να, να μιλήσει μαζί μας ή να κάνει κάποια ενημέρωση και ακόμα λιγότερο να μας δώσει κάποια ένδειξη των προθέσεών της σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. Εγώ τα μαθαίνω αυτά τα πράγματα μόνο πλαγίως και ανεπισήμως. Δεν με ικανοποιεί το να γίνεται μια τέτοια μορφή πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πλάγιο τρόπο και επισήμως να μην λέει τσιμουδιά η Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τους αξιωματούχους της ε, Κομισιόν που δώσανε αυτά τα στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να βασίζεται η διαμόρφωση της θέσης του Κοινοβουλίου σε τέτοιε μεθόδους. Νομίζω ότι αξίζουμε μια διαφορετική μεταχείριση από αυτή που μας επιφύλαξε η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ανδρέα Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσίασή του χαίρομαι γιατί μείνατε στο πλαίσιο στο οποίο είχε καταλήξει το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2013. Όμως, εγώ ανησυχώ, ανησυχώ για την αξιοπιστία του προτινομένου προϋπολογισμού. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια λάβαμε αιτήματα για περισσότερα χρήματα προς το τέλος του χρόνου κάθε φορά και για το 12 ξέρετε ότι ακόμα χρωστάμε και θα τα πρέπει να τα δώσουμε με τον φετινό προϋπολογισμό του 13. Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο προγραμματισμός του προϋπολογισμού. Στην παρουσίασή σας σταμάτησα σε αρκετά σημεία στα οποία δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο στις προβλέψεις σας, αλλά θα αναφερθώ μόνο σε δύο. Καταρχάς για τα ράλ. Είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι υπήρχε μια ισορροπία στο τέλος του χρόνου, ε, έμειναν μάλλον 200 εκατομμύρια από τα ράλ. Είπατε ότι εσείς ε, περιλαμβάνετε άλλα 70. Είστε σίγουρος για τα ποσά αυτά. δεν εγκαταλείπονται κάποια προγράμματα, κάποια άλλα προγράμματα δεν επιταχύνονται. Εν πάση περιπτώσει εγώ αμφισβητώ την αξιοπιστία των αριθμών αυτών στον προϋπολογισμό που προτείνεται. Θα έχουμε άλλα 130 δις δηλαδή για το 15 γιατί τον επόμενο χρόνο όλα τα ραλ που είχαμε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου θα πρέπει να διαγραφούν. Μπας περιπτώσει πρέπει να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Το δεύτερο το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι οι εξελίξεις των ταμείων συνοχής. Εσείς είπατε ότι για το 2013 έχετε 52 δις, ο προϋπολογισμός για το 2013 είναι 55 δις και ξαφνικά για το 2014 πέφτει στα 47 δις. Ξέρετε ότι η χρηματοδότηση της συνοχής δεν ακολουθεί τον ρυθμό, τον χρονικό της δημοσιονομικής διαδικασίας. Κάποιοι ξεκινούν προγράμματα σε διαφορετικές ημερομηνίε και συγχρηματοδοτούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οπότε πώς καταλήγεται σε αυτούς τους αριθμούς, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να μας εγγυηθείτε την αξιοπιστία των αριθμών που μας χρήνετε. Ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφοι, όλοι πήραν το λόγο και εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω δύο παρατηρήσεις και να θέσω ένα ερώτημα. Μία πρώτη παρατήρηση κύριε Επίτροπε σχετικά με την παρουσίαση του εγγράφου στην πρώτη σελίδα λέτε ότι στα πλαίσια των υποθέσεων εργασίας τις οποίες λάβατε υπόψη σας υπάρχει συμφωνία των τριών προέδρων της 6ης Μαΐου για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις της πολιετών δημοσιονομικών προβλέψεων επί τη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου και του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου. Γιατί είμαστε νομικά αυστηροί ή αναφερόμαστε γενικά σε πολιτικά έγγραφα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν έχουν καμία νομική αξία. Έχουν φυσικά ισχυρή πολιτική αξία. Και είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε υπόψη μας. Συνεπώς λοιπόν εμείς έχουμε το ψήφισμα της 13ης Μαΐου και μένουμε σε αυτό και πρέπει να το αναφέρετε. Αυτό είναι μια μικρή προειδοποίηση. Ε, μας έχει ενοχλήσει πρόσφατα η προσπάθεια να γίνονται κάποιες παρουσιάσεις και κάποια σχόλια ιδιαίτερα αισιόδοξα σε σχέση με την κατάσταση ε, την οποία βρισκόμαστε. Θα πρέπει και οι μεν και οι δε να είμαστε ιδιαίτερως επιφυλακτικοί πριν τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Μια δεύτερη παρατήρηση εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα, μετά από αυτά που άκουσα και από τους συναδέλφους. Εντυπωσιάζομαι και εγώ και όπως όλοι οι προηγούμενοι, σας ευχαριστώ για τους αριθμούς που μας δώσατε, είναι ξεκάθαροι και μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός του 14 θα μειωθεί ισχύρα σε σχέση με τον 13 και σε σχέση με αυτόν που ψηφίστηκε και θα γίνει αντικείμενο εκτέλεσης μέσα και από τους, διαρθρωτικούς, μέσα από τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα ανώτατα όρια ως έχουν και να το πω καλύτερα όπως προβλέπονται επί τη βάση της αποφάσεως του Οκτωβρίου. Μειώνονται τα ανώτατα όρια αλλά ταυτόχρονα αυτό εξηγείται και μέσω ενός άλλου φαινομένου το οποίο αναφέρθηκε από κάποιους συναδέλφους. Δηλαδή, για πολλές κοινοτικές πολιτικές και ιδιαίτερα για τις πιο ακριβές εισαγωγικά πολιτικές. Τις ενημερώνουμε, τις επανευρίσκουμε, εφευρίσκουμε αν θέλετε κάθε 7 χρόνια. Κάθε 7 χρόνια υπάρχει αν θέλετε μια ανάσα, ένα κενό. Και για κάποιους μήνες δεν μπορούμε να εργαστούμε γιατί υπάρχει ένα πραγματικό κενό και περιμένουμε τους καινούριου κανόνες για την κατάθεση των νέων ετοιμάτων και προγραμμάτων. Εάν λοιπόν αυτή η μείωση του ρυθμού που σημειώνεται ανά επταετία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γενικότερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα έλεγα εντάσσεται σε μια περίοδο εκτατική και πληθωριστική, εντάξει. Αλλά όμως τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Η στιγμή είναι πολύ κακή και το Συμβούλιο, ξέρετε, έχει προτείνει το Σύμφωνο Ανάπτυξης προσπαθώντας έτσι ώστε αυτά τα μικρά μέσα του μικρού κοινοτικού προϋπολογισμού να στηρίξουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν γίνεται αυτό η Ευρώπη βοηθάει ακόμα λιγότερο τη στιγμή που η Ευρώπη έχει ανάγκη βοήθειας. Λοιπόν, στην ουσία πρόκειται για ένα φαινόμενο, ένα συμβάν όπως λένε οι οικονομολόγοι, προκυκλικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό και νομίζω ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε στο να αμφισβητήσουμε τους ρυθμούς που ακολουθούμε και τις συνέπειες αυτές της ανακαίνησης και ανανέωσης των πολιτικών την ίδια στιγμή που ανανεώνουμε τη νομική βάση, τους ορίζοντες και τις προτεραιότητες όλων των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, να σας θέσω και ένα ερώτημα. Μετά και από τα ερωτήματα που έθεσαν ορισμένοι συνάδελφοι για τη διαχείριση των πιστώσεων πληρωμών για το 2013 και 2014. Εργαζόμεθα όλοι και όταν λέω όλοι αναφέρομαι σε εσά και σε εμά πάνω σε αυτό το θέμα θεωρώντας πρώτον ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το ταπ 2 για να αυξήσουμε κατά 11 δις 200 εκατομμύρια τις πιστώσεις πληρωμών του 2013 και δεύτερον ελπίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή θα καλύψει τα επιπλέον προβλήματα που αναδύονται το 2013. Ακόμα και αν συμβεί λοιπόν αυτό, θα υπάρξει το λεγόμενο backlog, ένα προηγούμενο όταν λέω θα λύσει τα προβλήματα του 2013, αναφέρομαι στα προβλήματα νομικής φύσεως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη νομική υποχρέωση να πληρώσει το 2013 όλων των αποδείξεων που θα κατατεθούν πριν από το τέλος του Οκτωβρίου. Ό,τι ακολουθήσει μπορεί να πληρωθεί τον επόμενο χρόνο. Και ήδη το 2013 στην αρχή του χρόνου η Κομισιόν πλήρωσε τα υπόλοιπα του 12 αλλά το 2013 κληρονόμησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πάρα πολλούς απλήρωτους λογαριασμούς από τον προηγούμενο χρόνο. Και φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Το τέλος δηλαδή του 2013 θα έχουμε υπόλοιπα απλήρωτα που θα επιβαρύνουν τις πιστώσεις πληρωμών του 2014. Τι σκοπεύετε να κάνετε εδώ με τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας τώρα που είναι προβλέψεις βέβαια αλλά παρόλα αυτά έχετε την δυνατότητα να προβλέπετε σωστά τα πράγματα και πώς προβλέπετε να συνδέετε εσείς το θέμα των πληρωμών του 13 με τις πληρωμές του 14. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, πολύ πλούσια συζήτηση. Ας ξεκινήσω με τις υποθέσεις για το 2013. Είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα συμβεί και έχει συμβεί το 2013 και δεν αναφέρομαι μόνο στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές νομικό σχέδιο αλλά και ε, στην διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού. Είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ ότι το ΕΚΟΦΗΝ σήμερα θα επιβεβαιώσει τη θέση της Κορεπέρ για την Κροατία. Έχει μεγάλη πολιτική σημασία αυτό, συμπολική σημασία, όπως κάναμε και πέρσι με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς, να ξεχωρίσουμε την υποδοχή στην Κροατία από ε, τα άλλα θέματα. Εγώ ε, γιορτάζω για δεύτερη φορά, γιόρτασα προσωπικά την προσχώρηση της ε, Πολωνίας το 2004 και τώρα ε, γιορτάζω την προσχώρηση της Κροατίας για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, είναι κάτι που γίνεται. Αυξάνουμε τις πιστώσεις ε, οι οροφές αυξάνονται κατά 374 εκατομμύρια ευρώ και καλώς. Τώρα, ως προς το σχέδιο προϋπολογισμού που ε, τροφοδοτεί τις πληρωμές για το 2013, αυτό δεν είναι σωστό. Είχαμε μια πολιτική απόφαση για τα 3,7, για τα 7,3 διορθώνει ο Επιτροπός, Αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρχει ρευστότητα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και για τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να έχουμε τέτοια δυνατότητα. Αλλά δεν τελειώνει η ιστορία εκεί. Και η κυρία Γένσεν και ο κύριος Μούλτερ, η Χέλκα, ο κύριος Σόουζα, ο Αλά, πολλοί το έθεσαν αυτό το ερώτημα για αυτά τα προβλήματα ε, ε, στο ετήσιο προϋπολογισμό. Τα 11,2 θα χρησιμοποιηθούν για τις νομικές υποχρεώσεις, προφανώς. Και κάτι που μπορεί να ξεφύγει μέχρι το τέλος της χρονιάς από τις πιστώσεις. Δεν μιλάω για τα ίδια νούμερα, γιατί τώρα οριστικοποιούμε τις τελικές εκταμιεύσεις για τα προβλήματα του 2012 Ευτυχώς τα έχουμε αφήσει αυτά πίσω μας. Εάν λοιπόν είναι κάτι το φυσιολογικό, έρχονται τα θέματα στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, προβλήματα εκ των υστέρων και έχουμε εκεί 5-6 δις. Αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει. Ίσως είναι λίγο παραπάνω από αυτό το ποσό. Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι να πληρώσουμε φέτος τους λογαριασμούς, τους νόμιμους, τους θεμητούς που έρχονται. Χρειαζόμαστε 11,2 δις φέτος για να μην μπούμε σε πραγματικά προβλήματα όχι μόνο πιστώσεων αλλά και ρευτότητα. Δεν είναι δηλαδή οι καθυστερημένοι λογαριασμοί που φτάνουν τον Εύριο το Δεκέμβριο το βασικό πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Στην παρουσίασή μου και για την Κροατία και για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 2 ε, τα έχω περιλάβει αυτά τα 11,2 δύο διαφορετικές υποθέσεις για το 2013 ε, στο οποίο νούμερο αναφερθήκατε πολύ ε, Υπάρχει και το πρόβλημα του σημείου αναφοράς. Φυσικά δεν είναι συνήθιση η διαδικασία αυτή. Φυσικά και έγινε επιλογή και έχω συζητήσει με πολλούς από εσάς το ζήτημα αυτό για το πώς θα παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός την επόμενη χρονιά. Ποιο θα είναι το σημείο αναφοράς που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχετε δίκιο. Τα συμπεράσματα είναι συμπεράσματα. Δεν είναι ένα νομοθέτημα που έχει ήδη εγκριθεί γιατί χρειάζεται η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Επιλογή μας λοιπόν ήταν να περιμένουμε, αλλά αυτό δεν είναι καλό για τη διαδικασία. Και επιλογή μας ήταν να αξιοποιήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων για να αλλάξουμε το προφίλ. Διότι θεωρούμε ότι έχει ολοκληρωθεί το της ε, ανεργίας των νέων και μπορεί να γίνει έμπρος φορτωσιακή. Υπάρχει σημαντική υποσημείωση σε κάθε σελίδα της εισαγωγής της παρουσίασής μας. Μένει να επιτευχθεί η συμφωνία και θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα αριθμητικά μας στοιχεία στη συμφωνία που θα επιτευχθεί μέσω μιας τροποποιητικής επιστολής την οποία μπορούμε να συντάξουμε μέχρι τη σύγκληση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Έχουμε αυτά τα περιθώρια. Έχουμε λοιπόν τη διπλή υπόθεση για το σημείο αναφοράς και έχουμε κάνει αυτές τις υποθέσεις πάνω στις οποίες έχουμε βασιστεί ε, για να ε, απεικονίσουμε και το πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και το ίδιο ισχύει και με τη νομική βάση. Που ήταν και το βασικό ερώτημα της ε, Σιδόνια και άλλων. Ε, αυτές τις υποθέσεις λοιπόν έχουμε και τα σημεία αναφορά. Πολλοί από εσά εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το επίπεδο του προϋπολογισμού. Φυσικά, ούτε εγώ είμαι ενθουσιώδης ε, με το προϋπολογισμό του 2014. Σίγουρα δεν υπάρχουν λόγοι ενθουσιασμού. Ο κύριος Χάρτ, ο κύριος Χάσχολτ και η κυρία Άντερσεν τάχθηκαν κάπως υπέρ αυτής της ε, εξοικονόμησης και περικοπών του κόστους για το 2014, κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τα λεγόμενα της ε, Σιδόνια του κυρίου Σόουζα. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό ήταν και το εγχείρημα στο οποίο είναι πλάκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με αυτό το οποίο είναι εφικτό, με αυτό το οποίο έχουμε. Και σαφέστατα δείχνει η προσπάθειά μας ε, το σημείο στο οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας. Εκεί όπου ε, φορτώνουμε με κονδύλια για να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα και εκεί που έχουμε όπιστο βαρύ προγραμματισμό. Τώρα, είναι και μεγάλη συζήτηση για τις εκταμιεύσεις για το 2014. Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει και με το, από το Σαλβαδόρ, τη Χάιντε, Χέλγκα κλπ. Νομίζω ότι γνωρίζετε τη λογική του πρώτου έτους μιας ε, προγραμματικής περίοδου ενός πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα έχουμε βραδία εκκίνηση σε τομείς όπου γίνεται sharp management στα διάφορα προγράμματα και σχέδια. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών. Χρειάζεται χρόνος και αυτή είναι η υπόθεση εργασίας σίγουρα για το Horizon 2020, για την έρευνα, για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό ρώτησε και η Χέλγκα άλλωστε. Όντως η ανάπτυξη της υπαίθρου ξεκινάει αργά. Ε, αργούν να ξεκινήσουν τα προγράμματα σε αυτό το τομέα. Για να καταλάβετε το πνεύμα του προπολογισμού του 2014 είναι απαραίτητο να κάνετε το διαχωρισμό μεταξύ των σχεδίων και project που μπαίνουν στο Sharp Management και των άλλων που ήδη μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης αρχής γενομένης από το 2014. Είναι περίεργη αυτή η σύνθεση των ε, πληρωμών και φαίνεται και στη διαφάνεια υπαριθμών 6, δεν ξέρω αν μπορούμε από τεχνικής πλευράς να την ξαναδείξουμε στην οθόνη, διότι φαίνεται ξεκάθαρα πόσο πρωτότυπη είναι η σύνθεση των πληρωμών στο πρώτο έτος ε, των δημοσιονομικών προοπτικών. Μόνο το 8% των ε, πληρωμών ή εκταμιεύσεων προέρχεται από νέες πιστώσεις την πρώτη χρονιά. Είτε μιλούμε για γεωργικές δαπάνες, είτε για οτιδήποτε άλλο, για δαπάνες διοίκησης. Και επομένως βασιζόμαστε σε αυτή τη ρεαλιστική υπόθεση εργασίας, ότι σε διάφορες κατηγορίες πληρώνουμε με τις εκρεμείς υποχρεώσεις και έχουμε το 1 τρίτο των ραλ, των υπολείπων προς εκαθάριση. Είναι περίεργη αυτή η ανάλυση του προϋπολογισμού και είναι κάτι που γίνεται μόνο την πρώτη χρονιά και τροποποιείται σε κάποιο βαθμό για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση κατά την άποψή μου και έχει σχέση και με τη σύνθεση των περιθωρίων. Έχετε δίκιο. Ε, δεν έχουμε περιθώρια ε, για τις πληρωμές. Και ο Σαλβαδόρ και ο κύριος Χάιντερ και ο Αλέν έθεσαν αυτό το ερώτημα. Έχουμε ένα περιθώριο 528 εκατομμυρίων ευρώ για τις πιστώσεις δεν είναι μεγάλο πράγματι. Είναι όμως ένας τρόπος να διαχειριστούμε καλύτερα τις προτεραιότητες που θα προκύψουν μετά τις αναγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι κάτι που εκφράστηκε επανειλημμένος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν ξεκινούμε με μεγάλα περιθώρια. Αυτό είναι η αλήθεια. Τα 500 όμως εκατομμύρια μας επιτρέπουν μια κάποια ευελιξία, όπως και αν χρησιμοποιηθούν τελικά. Μια κάποια κατανομή για την υπόλοιπη ε, περίοδο των ε, χρηματοδοτικών προοπτικών. Και έρχομαι στο πραγματικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Συνόδου και κατά πόσο θα λειτουργήσει η πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων σε σχέση με το εργαλείο αυτό που θα βοηθήσει για την επίλυση των προβλημάτων της νέας γενιάς στην Ευρώπη. Για να είμαστε ρεαλιστές, αρμοδιότητα κύρια έχουν τα κράτη-μέλη δεν μπορούμε εμείς να καλλιεργήσουμε υπερβολικές προσδοκίες. Έχουμε βασικά εργαλεία και χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις ενίοτε καθόλου δημοφιλείς ε, στην αγορά εργασίας. Και αυτά είναι όλα αρμοδιότητα και ευθύνη των κρατών μελών. Ώστε να, όμως προκειμένου αυτά να είναι αποτελεσματικά, λειτουργικά και βεβαίως δεν μπορώ να απαντήσω τώρα σε όλα τα ερωτήματα. Ε, έχουμε και το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε να πω ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ήδη έχει μπει στον κανονισμό για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επί τη βάση της πρότασής μας της 19ης Ιουνίου ζητήσαμε να συμπεριληφθεί αυτό ως νομική βάση το, ε, και στον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα πρέπει να υπάρξει νομική βάση. Δεν είναι όμως αυτό το βασικό ε, πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό που αναφέρατε εσείς, ο κύριος Χάσφορντ, ο κύριος Κόλμανε, και ο κύριος Μούλτερ, μεταξύ άλλων. Δηλαδή, είναι μια πολιτική δήλωση και μόνο ή είναι κάτι περισσότερο. Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά λειτουργικά, αποτελεσματικά. Η προπαρασκευαστική δουλειά για το 2014 πρέπει να ξεκινήσει από το 2013 επί τη βάση αυτών που γνωρίζουμε για το πώς θα πρέπει αυτό το εργαλείο να λειτουργήσει. Για μένα θα πρέπει να λειτουργήσει ώστε να προσφέρει το Youth Guarantee, ε, ε, κάτι το οποίο γίνεται στις σκανδιναβικές ε, χώρες. Εγγύηση στους νέους είτε για απασχόληση είτε για κατάρτιση. Δεν δουλεύει όμως στα 24 από τα 27 κρατη Για να γίνει λοιπόν λειτουργικό και αποτελεσματικό αυτό το εργαλείο έχουμε χρήματα με την έμπροσθεν φόρτωση. Και από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. 170 εκατομμύρια από την ενέργεια, από το Ταμείο Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, 640 από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και 400 περίπου κάτι εκατομμύρια από ε, το Connecting Europe και πάλι από άλλο σκέλος του. Αλλά όλα αυτά είναι γιατί τα project αυτά ξεκινούν αργά, καθυστερημένα. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δώσω νέες εγγυήσεις, ωστόσο θα ήταν εξαιρετική αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει του προγράμματος για την οικονομική ανάκαμψη να μην πετύχουμε με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Θα ήταν αποτυχία δηλαδή για την Ευρώπη να υιοθετήσει άλλη μια πρωτοβουλία χωρίς να έχει αντλήσει τα διδάγματα του προγράμματος της οικονομικής ανάπτυξης ανάκαμψης. Θα ήταν μια αποτυχία αν όλα αυτά παραμείνουν στη σφαίρα των πολιτικών ε, ε, ευχολογίων ή δηλώσεων. Και είναι, τέθηκε και το ερώτημα αυτό από τη Χέλγα. Κατά πόσο οι μειώσεις από κάποια προγράμματα μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν για τα συστήματα κοινής ανάληψης κινδύνου και συγχώνευσης δεν είναι μεγάλα τα ποσά για το πρώτη χρονιά, το 2014. Ε, η μόχλευση είναι ικανοποιητική και μπορούμε να, έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και το κόσμο και όλα με ορίζοντα το 2020. Είναι σταθερή η κατηγορία 4 στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Υπάρχει τώρα το θέμα της ε, μείωση των ποσών για την προενταξιακή βοήθεια, αλλά επειδή έρχεται η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια προενταξιακή χώρα. Τα άλλα στοιχεία αφορούν τις τεράστιες, τις υπεράνθρωπες προσπάθειές μας με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσουμε την Αραβική Άνοιξη. Τα τελευταία χρόνια αυτό ήταν μια θαυμάσια προσπάθεια που οδήγησε σε ενίσχυση των εργαλείων που έχουν να κάνουν με την Αραβική άνοιξη. Τώρα αν το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό ή όχι, αυτό είναι δική σας κρίση. Αλλά υπήρξε πράγματι μεγάλη ε, αύξηση των πόρων στον τομέα αυτό. Βέβαια υπάρχουν τώρα πολλά προγράμματα στα οποία υπάρχει τώρα χρηματοδότηση από πηγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε με τη φιλοσοφία περισσότερα με λιγότερα. Δεν χρειάζεται να περιμένει οι χώρες αυτές πιο πολλά α, κονδύλια. Στην κατηγορία 5. Αγαπητή μου κυρία Χολμάιερ. Δεν ήθελα να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ήθελα να σας πληγώσω. Και να δείξω τις αρμοδιότητες της αρχής του προϋπολογισμού. Χρησιμοποίησαμε τα δικά σας στοιχεία με τα τελευταία στοιχεία για το πάγωμα των αποδοχών των υπαλλήλων για το 2013-14 και 14 συγγνώμη, όλα αυτά συμφωνηθήκαν, αλλά δεν νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα. Αύριο, αύριο, ναι, ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι λοιπόν τα δικά σας στοιχεία εκτός από το τελευταίο αυτό στοιχείο του παγώματος των αποδοχών που βέβαια αλλάζει τις δικές σας ε, προβλέψεις εναντί των δικών μας προβλέψεων. Αλλά πρέπει να πω ότι λόγω σεβασμού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο εσείς δεν πήρατε την επιστολή μου. Όχι λέει κυρία Χολμάιρα εκτός μικροφώνου. Τα άλλα θεσμικά όργανα όχι μονάχα πήραν την επιστολή μου, έχουμε, έχουμε κάνει περικοπές και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχαμε κάποια περικοπή στα θέματα αυτά. Και δεν είχα καμία πρόθεση να σας προσ βάλω ή να προκαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε ένα θέμα με τις συντάξεις. Μέχρι τώρα είναι βιώσιμο το καθεστώς αυτό, αλλά εμεί καταστρέφουμε τώρα τις, στατιστικές, τις στατιστικές. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες σε επίπεδο διαχείρισης ιδίως των αποκεντρωμένων φορέων που βλέπω πόση μεγάλη δυσκολία έχουν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και δεν έχουν επαρκείς ανθρωπίνους πόρους. Μιλούσα με τον Μισελ Μπαρνιέ που νιώθει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού για τις εποπτικές αρχές, για τις χρηματαγορές. έλεγε και όλοι Ρεν, πόσους ανθρώπινους πόρους χρειάζεται για να ε, εκτιμήσει καλύτερα όχι μόνο το κρατικό χρέος αλλά και τις μακροοικονομικές ανισομέρειες στα 28 κρατημέλη. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν με την περικοπή των θέσεων στο οργανόγραμμα. Για τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν ξέρω. Ίσως υπάρχει μια μείωση του αριθμού των παιδιών. και στο επίπεδο των, της των συντάξεων υπάρχει πραγματικά η ανάγκη να είμαστε φιδωλοί. Στην κυρία Χέρτσοκ δεν θέλουμε να έχουμε διωγγωμένα ποσά στο ίτερ μέσα στον προϋπολογισμό, αλλά αν έχει γίνει αυτό, έχει γίνει από τα κράτη-μέλη και δεν πρέπει αυτό να υποσκάπτει άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. Κυρία Άντριασεν, δεν είναι πάντα τόσο μεγάλη αξιοπιστία του σχεδιασμού, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να ψηφίζει κανείς κονδύλια. Την προηγούμενη φορά είχατε επί... επικροτήσει την ανάγκη να είναι περιορισμένοι η προϋπολογισμοί, αλλά εδώ είναι η δυσκολία της διαφοράς μεταξύ του σχεδίου προϋπολογισμού και του τελικού αποτελέσματος που δεν μας επιτρέπει να έχουμε απόλυτα επακριβή σχεδίαση. Κύρια Χάουγκ. Ναι, πράγματι υπήρχε κάποιο λάθος στους πίνακες μας για το πρόγραμμα LIFE, όπως είπατε, για το 2014-2020. Είναι 3,1 δισεκατομμύρια, όχι 3,4 δισεκατομμύρια αλλά πολλές φορές αναφέρεται και το κόστος λειτουργίας και αλλού όχι και είναι δύσκολη η σύγκριση δύο ετών περιόδων. Αλλά δεν έχω τα λεπτομεριακά στοιχεία να σας απαντήσω. Πράγματι υπάρχει εδώ ένα λάθος. Ελπίζω ότι είναι μόνο ένα το λάθος στους πινακές μας. Το θέμα του τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Το ερώτημα του Γιάνν Μούλτερ. Η δική μου εντύπωση είναι η Ευρώπη είναι τόσο γεμάτη με προβλήματα και ερωτηματικά και αβεβαιότητες. Πρέπει να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα και όχι ένα αρνητικό μήνυμα στους λαούς της Ευρώπης. Γι' αυτό δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ ένα σενάριο μη συμφωνίας για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Θα είναι μαύρο σενάριο αυτό για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε το ταχύτερο δυνατόν μια συμφωνία για να προχωρήσουμε με τις νέες πρωτοβουλίες μας. Αλλά εξακολουθούν οι διαπραγματεύσεις τώρα. Δεν θέλω. Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα. Δεν πρέπει να δώσουμε αρνητικά μηνύματα, πρέπει να τονίσουμε την θετική πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γιατί η κατάσταση ήταν πιο δύσκολη σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις από ό,τι στο παρελθόν για τις προοπτικές 2007-2013 τότε που ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμα. Μπορούμε να σταματήσουμε λοιπόν εδώ τη συζήτηση. Και αυτό ήταν το τελικό μου σχόλιο. Ότι ο καιρός της Κασάνδρας έχει παρέλθει. Ελπίζουμε λοιπόν ότι δεν θα επαληθευτούν οι προσδοκίες οι προβλέψεις Κασάνδρας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας και για τις λεπτομεριακές απαντήσεις που κάνατε, που δώσατε για όλους τους ε, Ομιλούντε, Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μα και αύριο πρωί στην Επιτροπή προπολογισμών από τις 9 ω το 10.30 σε αυτή την ιδία αίθουσα. Και με την ευκαιρία αυτή θα προκύψει και η εντολή μας για τον τριμερή διάλογο προς τον εισηγητή μας για το 2014 τέλος τη συνεδρίασης.